Chers collègues, euh, bonjour. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σας. Να ξεκινήσουμε και πάλι τις εργασίες μας ε, αφού τη είχαμε αλλάξει χθε το βράδυ. Λοιπόν, ε, όπως σας είπα σήμερα, έχουμε αλλάξει τη σειρά ε, ανάμεσα στο 13 και στο 26 και τώρα το λόγο έχει η κυρία Σάρια Σαγιά για να μπορέσει να μας παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησης της ε, για τις δημογραφικές αλλαγές και τις συνέπειές τους στο μέλλον της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γνωμοδότησή μας που απευθύνεται στην, ε, περιφερειακή, στην Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής. Έχετε το λόγο, κυρία Σαγιά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα θυμάστε ότι στην ε, Επιτροπή μας εδώ ε, είχαμε εκπονήσει για τις δημογραφικές αλλαγές και μάλιστα το κ. Μάν ήταν συγητής, μια ε, σημαντική και λεπτομερή γνωμοδότηση. Τώρα συζητούμε τις επιπτώσεις των δημογραφικών αλλαγών στην μελλοντική πολιτική συνοχής. Όπως γνώριζετε, ε, μακροπρόθεσμα οι δημογραφικές αλλαγές θα δημιουργήσουν σημαντικές καινούριες προκλήσεις και απαιτήσει σε πολλές από τις ε, περιφέρειες των 27 χωρών και ενδεχομένως και οποιονδήποτε άλλων νέων χωρών ε, προσθεθούν μεταξύ. Οπότε η περιφερειακή πολιτική σε εθνικό και, κοιν, κοινοτικό επίπεδο θα πρέπει να προσαρμοστεί για να αντιμετωπίσει αυτές τις νέες προκλήσεις. Και τα τα ταμεία θα πρέπει να λάβουν υπόψη περισσότερο τις δημογραφικές αλλαγές. Οι περιφερειακές πολιτικές είναι κλειδί για τις περιφέρειες προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτές τις αλλαγές. Το 2007, μάλλον για την περίοδο 2007-2013, τα κράτη-μέλη σκοπεύουν να ε, δαπανίσουν πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ ε, σε μέτρα ε, για δημογραφικά ε, προβλήματα. <clears throat> Θα ε, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και διαφορές ε, στο κατακεφαλήν ΑΕΠ ε, στην κατανομή των ποσών ανάμεσα στις περιφέρειες. Και αυτό είναι το βασικό μήνυμα της νομοδότησής μας, ότι το ΑΕΠ είναι ένας καλός δείκτης, βέβαια χρειαζόμαστε και άλλους δείκτες. Και όταν, έχουμε, όταν συζητάμε το θέμα των δημογραφικών αλλαγών, θα πρέπει να εξετάζουμε και άλλους δείκτες στις περιοχές όπου η, ε, η γύρανση θα είναι πιο γρήγορη, ε, αυτές οι περιοχές ε, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως περιοχές δοκιμής. Προκειμένου εκεί να αναζητήσουμε καταρχήν την λύση των προβλημάτων. Οι καινοτομίε που θα δοκιμαστούν εκεί θα πρέπει να αφορούν πολλούς τομείς. Για παράδειγμα, αύξηση τη παραγωγικότητα στον τομέα μέρημνα και περίθαλψη για του ηλικιωμένου με τη χρήση τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Επίση, ε, προσπάθεια να περιμένουν οι ηλικιωμένοι υγιεί, δραστήριοι και ικανοί να ζουν στο σπίτι. Αυτά είναι, είναι, αυτές είναι δύο από τι περιοχέ όπου οι καινοτομίε θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Λαμβάνοντα υπόψη ότι η Κομισιόν έχει ήδη ξεκινήσει μια πιλωτική συνεργασία ε, στον τομέα της δραστήριας και υγιούς γύρανσης. Ε, στην γνωμοδότησή μα θα μπορούσαμε ε, να συμπεριλάβουμε αυτά τα δύο θέματα και να τα υπογραμμίσουμε, να υπογραμμίσουμε την ανάγκη δηλαδή τέτοιου είδους πιλωτικών project. Στη μελλοντική πολιτική συνοχή χρειαζόμαστε λιγότερη γραφειοκρατία και θα πρέπει να προσαρμόζεται στα, στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων με επικέντρωση στην παραγωγικότητα, την ε, απασχόληση και άλλους στόχους της πολιτικής της Ευρώπη 2020. Μην ξεχνάμε ότι καινοτομίες δεν χρησιμοποιούνται αυτές καθ' αυτέ, ε, δεν είναι αυτός σκοπό Χρειαζόμαστε τις καινοτομίε για να λύσουμε τα κύρια προβλήματα των κοινωνιών μας, για παράδειγμα την γύρανση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα ακούσω και την γνώμη των ε, σκιωδών εισηγητών για αυτή την ομοδότηση και περιμένω να συνεργαστούμε ε, στο μέλλον. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για να δούμε τώρα ποιος επιθυμεί να λάβει το λόγο. li Η κυρία Λίν, επιτέλους κάποιος. Ευχαριστώ. Έχω κάποιες ερωτήσεις για το 12 και για το 17. Μιλάτε για την ενίσχυση της πολιτικής συνοχής. Υπό ποια έννοια θέλετε να ενισχυθεί. Επίσης το 21 αναφέρει ανακατανομές του προϋπολογισμού. Θα μπορούσατε να το διευκρινίσετε και σε αυτό το σημείο τι εννοείτε. Α, κάνω λάθος για τα διορθωτικά ταμεία. Κάνω λάθος στο έγγραφο. Euh, Για την εισηγήτρια. Δηλαδή η άποψή της πώς βλέπει αυτή την εξέλιξη, αυτό που μας ενδιαφέρει άμεσα και το αναφέρεται στην παράγραφο 3. Τι γίνεται δηλαδή, με ποιο τρόπο θεωρείτε, νομίζετε ότι θα αυτό το θέμα το δημογραφικό θα ληφθεί υπόψη και για ένα πληθυσμό που γυράσκει συνεχώς ε, παρόλο που αυτό δεν ενδιαφέρεται τουλάχιστον σαν κύριο στόχο για τον πληθυσμό αυτό από τη στιγμή που αποχωρεί από την αγορά εργασίας. Πρόκειται όμως και για μια πρόκληση για τους νέους. Έχουμε μια τεράστια διάφορα δύσκολη, το είπαμε και εδώ πέρα είπαμε ότι δυσκολεύονται να μπουν στην αγορά εργασίας και υπάρχουν όλο ένα και περισσότερο ηλικιωμένα άτομα. Κατά την άποψή μας πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή πέρα από μια διαπίστωση ότι ε, θα είναι περισσότεροι μιας κάποιας ηλικίας άτομα και σε σχέση με αυτό που έχει αναλάβει η κυρία Ομερόιτεν. Και εδώ για το ΕΦΣΕ υπάρχει ένα, ένας ρόλος που θα πρέπει να παίξει την προσαρμογή για το κοινωνικό ταμείο, δηλαδή ε, για το ε, εργασία, κοιτάζουμε ποια είναι η ηλικία. Όχι, δεν με διακατέχει η ιστερία για το πώς θα πρέπει να αποχωρήσει κανείς στα 60 χρόνια να συνταξιωτηθεί αλλά αν δεν προσαρμοστεί η κατάσταση με τις εργασίες πέρα από τα 60 χρόνια, δεν θα έχουμε τότε στη διάθεσή μας τα μέσα για να απασχοληθεί κόσμος ε, και από ηλικιωμένα άτομα. Και πέρα από αυτή την εξέλιξη δημογραφική, τουλάχιστον για τη δική μας την περίπτωση το κοινωνικό ταμείο, γιατί και το ε, περιφερειακό ε, ασχολείται, αλλά ε, υπάρχει και άλλη διάσταση, δηλαδή θα πρέπει να δούμε τι κόστος συνεπάγεται αυτό όπως αναφέρεται. Η κυρία Μωρέν επιθυμεί να λάβει το λόγο. Μήπως υπάρχει κι άλλος που επιθυμεί να λάβει το λόγο επίσης. Κύριε Μωρέν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ απόλυτα συμμερίζομαι τα όσα είπατε εσείς. Θα ήθελα τώρα να προσθέσω και κάτι άλλο που κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή γεωγραφικά, πώς κατανέμονται αυτές οι γεωγραφικές ε, ομάδες. Βλέπουμε την κάποια τάση που υπάρχει ο ηλικιωμένος πληθυσμός να είναι αγροτικός κυρίως και εδώ μπαίνουμε σε άλλα χωράφια, δηλαδή στο θέμα της πολιτικής συνοχής, γιατί δημιουργείται ένα διπλό πρόβλημα. Να δούμε πρώτα απ' όλα τι γίνεται εάν συμφωνήσουμε με την παρατήρηση της κυρίας Μπέρες ε, σε αγροτικό περιβάλλον ε, ποιες θέσεις απασχόλησης για τα άτομα ή γυράσκοντα άτομα τι θα γίνει και επίσης ε, για τη συνοχή την εδαφική ανάμεσα σε παρόμοιες δημογραφικές ομάδες ε, που γεωγραφικά έχουν διαφορετική καταγωγή ανάμεσα σε αστικό και σε αγροτικό περιβάλλον. Ο Πρόεδρος, κάποιος άλλος μήπως θα επιθυμούσε να λάβει το λόγο τώρα. Δεν βλέπω. Έχετε το λόγο κυρία μου. Ε, πολύ σωστά τα σχόλια αυτά. Ε, δεν είχαμε και πολύ χώρο για να καλύψουμε όλα αυτά τα θέματα σε αυτή την ε, λιτή μα νομοδότηση. Μπορούμε όμως να κάνουμε τροποποίησεις για το κοινωνικό ταμείο το οποίο ανέφερε η Πρόεδρος. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους πόρους για να ε, βοηθήσουμε την γυράσκουσα, το γυράσκο μας δυναμικό και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που χάνουν την εργασία τους λίγο πριν τη συνταξιοδότησή τους. Αυτοί είναι πολύ δύσκολο να ξαναμπούν ε, στην αγορά εργασίας, να ξαναρχίσουν να δουλεύουν, να βρουν μια θέση εργασίας. Οπότε ένα τμήμα των πόρων μας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να τους βοηθήσουμε αυτούς τους άνεργους ε, ηλικιωμένους. Ελίζαμπεθ, ε, για την διαφορά ανάμεσα ε, στις πόλεις αστικές δηλαδή περιοχές και τις περιοχές υπαίθρου. Πολύ σωστά ε, οι δημογραφικές ε, αλλαγές ε, θα γίνουν πιο σαφείς και πιο γρήγορα στη Βόρεια Σκανδιναβία, στην Ανατολική Γερμανία και στη Βόρεια Ιταλία. Αυτές είναι οι τρεις περιοχές της Ευρώπης που, πιο, που γυράσκουν πιο γρήγορα σε όλη την Ευρώπη. Οι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πολλές διαφορές ανάμεσα σε περιφέρειες. Αυτό είναι αλήθεια. Euh, Η Πρόεδρος, να ευχαριστήσουμε την εισηγητριά μας. Προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Αυτή ισχύει, μάλλον τώρα από τώρα. Ισχύει και θα είναι μέχρι τις 11 ε, Φεβρουαρίου στις 12 η ώρα το μεσημέρι και 15-16 Φεβρουαρίου συζητήσεις σχετικά με αυτό και θα, θα συζητηθούν και θα υιοθετηθούν ε, τον Απρίλιο 13-14 ε, Απριλίου ακριβώς γιατί η Περιφερειακή Πολιτική, η Επιτροπή αυτή θα πρέπει το Μάιο να ψηφίσει για την έκθεσή της επί και έτσι έχουμε κάποιο χρονικό διάστημα στη διάθεσή μας για να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Τώρα πριν να ψηφίσουμε να σας ε, κάνω μερικές ανακοινώσεις. Είπα χθε ότι θα είχαμε τη νέα κατανομή αρμοδιοτήτων, ότι θα σας ε, την ανακοινώσουμε ακριβώς ε, στη Γενική, για τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης ε, και ήδη έγινε μια ανακοίνωση αυτής της πληροφορίας με mail της 13 του Ιανουαρίου. Δεν θα υπάρξει μια νέα κατανομή, μια νέα διανομή αυτού. Σήμερα και για αν θέλετε να θα απαντήσετε κάτι, δεν το κάνετε μέσω mail και πάλι. Τώρα σχετικά με την σημερινή απογευματινή συζήτηση για τις συμβιβαστικές τροπολογίες για την έκθεση της κυρίας Όμερ Ρόιτεν που είναι στο σημείο 27 της σημερινής μας διάταξης. Είχα φράσει την επιθυμία από σήμερα ήδη να γίνει μια ανακοίνωση των συμβαστικών τροπολογιών, τις οποίες διαπραγματευόμαστε και η κυρία Όιμεν Ρόιτερ στις 10 σήμερα το πρωί θα έλθει σε διαπραγματεύσεις με ορισμένες πολιτικές ομάδες. Άρα λοιπόν μόνο στην αρχή του απογεύματος ε, θα έχετε στο χαρτί τυπωμένες αυτές τις ε, συμβασικές τροπολογίες, αλλά κατέλαβε βέβαια από τη στιγμή που θα τις διανύμουμε αυτές ε, τυπωμένες στο χαρτί θα μπορούν και να μεταβαστούν σε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους σας, ώστε όλοι να τα έχετε αυτά ακριβώς τη στιγμή που θα διεξαχθεί η συνάντηση και ανάμεσα στο ξεκίνημα σήμερα το απόγευμα και ζήτηση να μπορεί κανείς να τα μελετήσει και να τα συζητήσει στη συνέχεια. Και στο τέλος της απογευματικής συνάντησης ε, θα ξεκουραστούμε και κάπως ε, ευχάριστη στιγμή για να ευχηθούμε στον άλλο καλή χρονιά 2011. Δυστυχώς ο Επίτροπος δεν θα μπορέσει να παραστεί είναι στο Ντάβος με τους ε, μεγάλους του χρήματος, ε, του δημοσιονομικού συστήματος και εντάξει καταλαβαίνετε λοιπόν ε, θα έχουμε την ευκαιρία πάντως να έρθουμε σε επαφή με το Γενικό Διευθυντή Απασχόλησης του κ. Μπερβερή που θα είναι η τελευταία του συμμετοχή σε εργασίες μας παρόλο που θα γίνει άτυπα νομίζω όμως ότι σημαντικό είναι να χαιρετήσουμε την παρουσία του εδώ γιατί συνεργαστήκαμε πολύ καλά μαζί του όλα αυτά τα χρόνια. Να έλθουμε τώρα στο σημείο 14 της ημερήσιας διάταξης. Τι θα κάνουμε, θα ψηφίσουμε. Θα ψηφίσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης. Ε, λοιπόν, σχέδιο γνωμοδότηση της κυρίας Νάντια Ήρσα έχει να κάνει με την ισότητα γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Ένας από του σοσιαλιστέ δεν έχει φέρει την καρτούλα του για την ψηφοφορία. Όλοι οι υπόλοιποι... Παράγραφος 1. Τι έχουμε εκεί, δύο τροπολογίες. Τροπολογία 1 της κυρίας Στάιρακ, Εύελεν Ρενιέ, Έντιτε Ψηφίζουμε υπέρ. κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Και αν ψήφισαν όλοι, πέρασε ψηφοφορίας. 17 απορρίπτεται. Προχωράμε δύο τροπολογία κρήτου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά από την 1 έχουμε την τροπολογία 3, κυρία Σεστρέλα και Στάνακ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 4, Λόπες, μπουπάκη, ε, υπέρ κατά αποχές Κανονικά εγκρίνεται, αλλά για να δούμε, για να ελέγξουμε. Ξεκινάει η ψηφοφορία, παρακαλώ. Και αν ψήφισαν όλοι, πέρασε ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, έτσι. Πώ τι. Ναι, αλλά για να ψηφίσετε πρέπει να πατήσετε το κουμπάκι σας. Λειτουργεί η καρτούλα σας. Βάλτε το χεράκι σας μέσα, πιέστε και θα ψηφίσετε. Πέρα ψηφοφορία 20 υπέρ, 12 κατά, η αποχημία εγκρίνεται λοιπόν. Τροπολογία 5, Ροντζούλη υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2, συμβαστική τροπολογία α. Αρκετοί την προτείνουν, τουλάχιστον από δύο πολιτικές ομάδες, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Με την το 2 έχουμε τροπολογία 12, Εστρέλα και Σάνδρακ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 14, και Ρονζόλη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15, Ρονζόλη, Υπέρκατά κατά αποχές εγκρίνεται, παράγραφος 3, τροπολογία συμβαστική από τους εισηγήτρια πρώτα και μετά την σοσιαλιστική ομάδα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 3 και τροπολογία 19 μετά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 της Ρονσούλη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 Λοπές Φοντανιέπ και κ. Πουπάκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 απλών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Παραφό 4 τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές Τροπολογίε τροπολογίες 26-27 καταπίπτουν ψηφίζουμε 28 του σκοτωτού που μπορεί να συνδυαστεί με τις υπόλοιπες η συγκεκριμένη υπέρ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 4 και τροπολογία 29 της κ. Φιγκερέιντο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 Ρονζούλη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 Στάινρακ Εστρέλα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 Φιγκερέιντο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 34 Στάινρακ και Εστρέλα Εκεί μας έχουν ζητήσει προφορική τροπολογία, η κυρία Στάιρακ ακριβώς και η συγγήτρια ίδια, για την αρχή της τροπολογία που λέει calls on the member states to review the taxation κλπ. Καλύτερα κρατημέλη και κάποιος κάτι όχι, ψηφίζουμε έτσι τροποποιημένη 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35, Βιερστράινρεκ Ρεϊνιέ Εστρέλα, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος τώρα 5, τροπολογία 36, ψηφίζουμε υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 39, της κ. Κορνέλησεν, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 38 κατά πίπτη. ψηφίζουμε 37, του που συνδυάζεται με τις υπόλοιπε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5, τροπολογία 40, υπέρ κατά αμφίβολο, κανονικά εγκρίνεται. Θέλετε να το ελέγξουμε. Άντε, άντε να το ελέγξουμε. 40, ψηφίζουμε τη 40 παρακαλώ. Και αν ψήφισαν όλοι, πέρασε ψηφοφορίες 27 υπέρ, 11 κατά. Ναι, εγκρίνεται. 41 κορνέλες εν υπέρ. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, ελέγχουμε. Και αν ψήφισαν όλοι, πέρα στις ψηφοφορίες. 23 υπέρ, 16 κατά. Εγκρίνεται. Παράγραφος 6 τώρα, 45 της συγκήτριας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 47 καταπίπτει. Και τι γίνεται με τις υπόλοιπες, ναι, νομίζω ότι στέκουν με τις υπόλοιπες. Λοιπόν, 46 κρετού υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 44 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 48 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παραφώς 6, τροπολογία 49, φιγκερέιντο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 50 της κυρίας Ρονσούλη, Α, μια παρατήρηση από πλευρά τη συγκητρίας. Και από την ίδια τη συντάκτρια της τροπολογίας. Τροπολογία 50, μιλάμε για την 50, υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 52 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 51. Στάνερκ και Στρέλα υπέρ κατά αποχές γκρίνεται 53 Thomas Mann υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 φιγκερέιντο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 της ίδιας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 Φιγκρέντο και πάλι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 Thomas Mann υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 φιγκερέιντο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 φιγκερέιντο και πάλι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 φιγκερέιντο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 φιγκερέιντο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 7. Τροπολογία 64 για διαγραφή ψηφίσμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική λύση τώρα γάμα από δύο ομάδες, από τους φιλελεύθερους και τους σοσιαλιστές υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παραγραφό 7 που πάμε τώρα στην τροπολογία 67 της εισηγήτριας. Εκεί θα έχουμε πρώτα το σύνολο της παραγράφου που θα ψηφιστεί χωρίς το voluntary. Υπέρ λοιπόν του συνόλου της 67 χωρίς με το voluntary. Υπέρ. Το σύνολο της 67 είπαμε, χωρίς την λέξη voluntary. το σύνολο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αυτό χωρίς το voluntary. Ποιος είναι υπέρ του να συμπεριληφθεί και η λέξη voluntary. Κατά. Αντίθετη στο με τη διάθεσή μας. λοιπόν, για να δούμε, τους ελέγχουμε για να μπει αυτό το voluntary. Ah oui, oui, oui. <laughs> Tout le monde a pu voter, le vote clos. Και αν ψήφισαν όλοι, πέρας ψηφοφορίας, 25-17, άρα... Α, η αποχή, μία αποχή. Α, λοιπόν, ναι, με τη διάθεσή μας είχαμε με την καλή διάθεση, εντάξει, ευπρόσδεκτη αυτή, Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο της νομοδότησης αυτής, ηλεκτρονική ψηφοφορία, ξεκινάει η ψηφοφορία. Εντάξει, μυστική ψηφοφορία, ε. Για προσέξτε το αυτό. Και μην κάνετε λάθος και στο κουμπάκι που θα πιέσετε. Και αν ψήφισαν όλοι, πέρας ψηφοφορίας. Υπέρ 40, ένας Αντίθετος, οι αποχές δύο συγχαρτήρια στην εισηγητρία μας. Ε, Au point 15, ε, stratégie. 15, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωση ε, για την ασωμάτωση των Ρώμα. Ψηφίζουμε την Ρωμά της κυρίας Κίνγκα Γκάνς. Να σας υπενθυμίσω κάτι. Εκεί είμαστε στα πλαίσια ενισχυμένης συνεργασίας με την ε, Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών. Και τώρα Τροπολογία 1. Μπεναμιάς υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 του ίδιου συντάκτη εγκρίνεται. Πρώτη συμβαστική τροπολογία της εισηγήτριας και της κυρίας Παπαδοπούλου. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Στην παράγραφο 1, τροπολογία 5, να διαγραφεί Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία Β. Από δύο πολιτικές ομάδες. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μετά τροπολογία 8 για την παράγραφο 1α. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 4 του κυρίου Γκουρεάνου, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 2, συμβαστική τροπολογία Γ. Από τέσσερι πολιτικέ ομάδε. ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 14 της κυρίας Παπαδοπούλου. Α, κατα, καταπίπτει και αυτή. Στην παράγραφο 3, συμβιβαστική τροπολογία Δέλτα της εισηγήτριας. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 3, συμβιβαστική τροπολογία ε, από τέσσερις πολιτικές ομάδες, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 20 είναι μη αποδεκτή και μετά τροπολογία 21 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την τροπολογία 3, συμβαστική τροπολογία F, σίγμα ταφ, από τρεις πολιτικές ομάδες, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 3, ψηφίζουμε για την τροπολογία 23, σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα της τροπολογίας ψηφίζουμε πρώτα μέχρι το combat phenomenon, ψήφι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά, αποχές, νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα της τροπολογίας 23. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τις ψηφοφορία. 23 υπέρ, 19 κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται όντω. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 3 και πάλι, τροπολογία 24 της κυρίας Ιώτοβα. Ψήφι υπέρ. Μάλλον καταπίπτει. Τροπολογία 26 έχει αποσυρθεί. Συμβαστική ε, τροπολογία G από τέσσερις ομάδες ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι επόμενες και περνάμε στην παράγραφο 6. Συμβιβαστική τροπολογία H, ψήφι υπέρ, για την παράγραφο 6. Συμβιβαστική τροπολογία H, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προς την κυρία Ισηγητή, έχω μια ερώτηση. Στην παράγραφο 6. Συγγνώμη, συγγνώμη, στην παράγραφο 5. Α, όχι. Ζητώ συγγνώμη, αλλά ξεχάσαμε να ψηφίσουμε την παράγραφο 5. Τρει τροπολογίες που νόμιζα ότι καλύπτονται από τη συμβαστική λύση, αλλά δεν καλύπτονται. Στην παράγραφο 5 πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 37 για να, για να διαγραφεί το κείμενο. Ποιο είναι υπέρ τη τροπολογίας 37. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Τροπολογία 38. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 39. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Για την παράγραφο 5 έχουμε εγκρίνει λοιπόν την τροπολογία 39. Και επιστρέφουμε στην παράγραφο 7 τώρα. Συμβαστική τροπολογία I, Ι, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Παράγραφος 8 τώρα, τροπολογία 50. Ψηφί υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 49. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία J. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μετά την τροπολογία 8, τροπολογία 52. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 9. Α, συγγνώμη. Απορρίπτεται. Παράγραφος 9. Συμβαστική τροπολογία Κ. Από πέντε πολιτικές ομάδες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 9 έχουμε μια συμβαστική τροπολογία L, λάμδα, δύο ομάδων υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Στην παράγραφο 10 συμβαστική τροπολογία μη υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 10, τροπολογία 61, για μια νέα παράγραφο, τροπολογία 61, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 65 καταπίπτει. Μετά την παράγραφο 10, τροπολογία 68 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 11, Τροπολογία 70, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 71, πάλι Ουγγουράνου, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 11 και πάλι συμβαστική τροπολογία εν, νη, τριών πολιτικών ομάδων, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 12, τροπολογία 75, Μπαλντασάρε, ψήφι υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. Να το επαληθεύσουμε για την 75 άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Πολλές ψήφοι για το ΕΛΚ. Θα αφαιρέσω μία ψήφο. Ή θέλει κάποιος από το ΕΛΚ να αποσύρει μια ψήφο. Ωραία. Πέρασε η ψηφοφορία. 19 υπέρ, 24 κατά. Απορρίπτεται λοιπόν. Τροπολογία 76 καταπίπτει. Να ψηφίσουμε τη συμβαστική τροπολογία, μάλλον την τροπολογία 77 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται και τροπολογία όμικρον σοσιαλιστικής ομάδας ψηφί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 12 τροπολογία 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στην παράγραφο 13 καταπίπτουν οι τροπολογίες από, ε, λόγω της συμβαστικής νη. Μετά 85 της κυρίας Ασταγιά υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 14, 87 του κυρίου Γκουρεάνου υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 88 ψηφί υπέρ. δεν χρειάζεται. 88 Παραλαμβάνουμε υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 89 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 14, α, όχι, εγκρίνεται, λάθος, λάθος το είπα, 89 εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 14, τροπολογία 90 του κυρίου Μπαλτασάρα, μετά από μια προφορική τροπολογία για τη διαγραφή κάποιων λέξεων από το devise and adopt μέχρι το social welfare system. Διαφωνεί κανείς για την προφορική τροπολογία. Κάποιος διαφωνεί με την προφορική τροπολογία. Άρα δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την προφορική τροπολογία. Θέλετε να οργανώσετε μια φορά κατ' εξαίρεση. Όχι. Θα ψηφίσουμε λοιπόν ολόκληρη την τροπολογία 90 του κυρίου Μπαλτασάρε. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το επαληθεύσουμε για την τροπολογία 90. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. 23 υπέρ, 21 κατά εγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά υπέρ. Μετά την παράγραφο 15 περνάμε στην τροπολογία 95 όπου υπάρχει και πάλι μια προφορική τροπολογία να προσθεθεί η λέξη social. Δεν διαφωνεί κανείς για την προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε την 95 λοιπόν, όπως τροποποιήθηκε με την προφορική τροπολογία. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 96 και 97 δεν είναι παραδεκτές. Ψηφίζουμε λοιπόν για το σύνολο του κειμένου με ηλεκτρονική ψηφοφορία. on a pu. Et le, le PPE euh, essaie de Εντάξει και η ψήφη του ΕΛΚ. Βγαίνουν παραπάνω, αλλά αυτοπιθαρχείτε και μετά διορθώνετε το αποτέλεσμα. Λοιπόν, 43 υπέρ, μία ψήφος κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια προς την εισηγήτρια, την κυρία Κόντς. Αλλά έχει πάει και έχει κρυφτεί στο βάθο η συγκεκριμένη δεν ξέρω γιατί. Euh, Ωραία. Περνάμε στο σημείο 16. Τελειώσαμε δηλαδή με τις πληροφορίε. Στο σημείο 16 πλέον έχουμε Έχουμε τη γνωμότητα του κ. Μπαλτασάρ για την, προς την ε, Επιτροπή ΙΜΚΟ. Ενιά αγορά για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη. Είναι η πρώτη από τρεις νομοδοτήσεις. Είναι ε, παρακαλώ, ήσυχα εγκαταλείψτε την αίθουσα όσοι θέλετε να φύγετε. Baldassar, est-ce que je peux vous demander... Κύριε Βαλτάσαρ, μπορείτε να μας παρουσιάσετε την ε, γνωμοδότησή σας. Can you please be silent? It's not possible to work in these conditions. Ε, δεν μπορούμε να δουλέψουμε έτσι. Σας παρακαλώ πολύ λίγη ησυχία. Κύριε Βαλτάσαρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή είναι η αγορά είναι από τους ακρογωνιαίους λίθους ε, στο σχέδιο ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν, να το σκεφτούμε, πάνω από 20 εκατομμύρια επιχειρήσεις με 175 εκατομμύρια θέσεις εργασίας που προσφέρουν. Βέβαια, δεν σημαίνει αυτό το πράγμα ότι ο πλούτος ε, και η αύξηση του ΑΕΠ ε, πέφτει στους ώμους ε, της επιχείρησης και στα κέρδη της επιχείρησης. Αντίθετα όμως, ένα κανόνικο κοινωνικό σύστημα θέση εργασίας και ανταγωνιστική μισθή αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις που σίγουρα ακριβώς απαιτούνται για αρμονική ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας της ευρωπαϊκής αγοράς. Η σημασία αυτής της επιχείρησης είναι ότι και της πράξης αυτής είναι ότι θέλουν να προσφέρουν απαντήσεις στην ενιαία αγορά για καλύτερη πρόσβαση, συμμετοχή στην αγορά όλων αυτών των φορέων, των παραγόντων και των καταναλωτών και των εργαζομένων. Για να πετύχει κανείς αυτό το στόχο, τα μέτρα εδώ σε αυτή την πράξη αφορούν τέσσερις κύριους στόχους ε, υποστήριξης της επιχειρήσης ε, και διευκολύνοντας ε, την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την κοινωνική οικονομία μέσω συστημάτων που στοχεύουν σε αυτή τη βοήθεια, την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και τη χρησιμοποίηση όλου του δυναμικού του μαζί με τις ανάγκες των καταναλωτών και σε σχέση με τους νόμους αγοράς, τις ρυθμίσεις αγοράς και επίσης ρυθμίσεις για επαγγελματική κατάρτιση ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν σε αυτήν την αγορά οι εργαζόμενοι. Μετά από όλα αυτά, εντάξει, εγώ είμαι αρκετά ικανοποιημένο από το κείμενο, το έγγραφο αυτό πάνω στο οποίο θα χρειαστεί να ψηφίσουμε. Και θέλεις ακριβώ τη γνωμοδότησή μου να τονίσω ορισμένε πτυχέ που κατά την άποψή μου αποτελούν προποθέσει ε, απαραίτητε για τι εφαρμογέ αυτέ για την ανάπτυξη τη εσωτερική αγορά. Ειδικότερα αναφέρομαι σε διάφορε πτυχέ που εμεί τονίσαμε στην ε, έκθεση για την καλύτερη πρόσβαση ακριβώς της μικρών μεσαίων επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά με μείωση των υποχρεώσεων διοικητικού χαρακτήρα και επίσης αφαιρώντας οποιοδήποτε εμπόδιο κυρίως ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου έχουμε μια ανάπτυξη της τάξης του 26% στα κράτη-μέλη ψηφιακού εμπορίου και 17% πάει όταν έχουμε διαμεθοριακές ή ε, διακρατικές επαφές ε, και ε, να διευκολύνουμε στην κεφαλαγορά την πρόσβαση αυτών των εταιριών σε περίοδο κρίσης για πιστώσεις για τις επιχειρήσεις αυτές, ε, γιατί διαφορετικά αντιμετωπίζουν δυσκολίες να παραμείνουν στην αγορά και να εργαστούν όπως πρέπει και επίσης ε, τους δημόσιους διαγωνισμούς και προκηρύξεις να του χρησιμοποιήσουμε υπέρ τη κοινωνική ανάπτυξη. Και ακόμα τελικά έχει σημασία κάθε στήριξη σε αυτές τις επιχειρήσεις ε, και κυρίως τις μικρές ε, θα πρέπει να έχει να κάνει με τον κατάλληλο χώρο και να ευθυγραμμιστεί με την ε, Ευρωπαϊκή Στρατηγική του 2020. Μόνο συνδυάζοντα αυτό την υποστήριξη αυτέ τι επιχειρήσει με του κοινικού στόχου και του στόχου τη απασχόληση, έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε τον πραγματικό στόχο τη πράξη. Δηλαδή για μια κοινωνική οικονομία τη αγορά που να βασίζεται στην ανάπτυξη, στον ανταγωνισμό και στην κοινωνική πρόοδο. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ποιο θέλει να πάρει το λόγο. Κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύμφωνο με τον εισηγητή. Η εσωτερική αγορά είναι ακρογωνίως λίθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενιαία αγορά Δυστυχώς όμως έχει γίνει αρνητική έννοια στα μάτια των πολιτών μας. Γιατί έπαψε να είναι καινοτόμα, έπαψε να είναι μια ιδέα φρέσκια. Όμως η ενιαία αγορά καλύπτει και θέματα που δεν είναι οικονομικά. Κατάρτιση, ανταλλαγές διαφόρων τύπων, διαβίου, εκπαίδευση κλπ. κλπ. Εμείς περιμέναμε πιο πολλά θετικά στιγμιά στην πρόταση της Κομισιόν. Για παράδειγμα, θα θέλαμε να είχε υποβάλει Κομισιόν νομοθετικές προτάσεις για τις ε, υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος και για τις υπηρεσίες γενικού κοινωνικού ενδιαφέροντος. Η Κομισιόν Παλιότερα έλεγε ότι δεν είχε νομική βάση για να υποβάλει τέτοιου είδου νομοθετικέ προτάξει. Τώρα όμω με την συνθήκη τη Λισαβόνα υπάρχει αυτή η νομική βάση. Δυστυχώ όμω η Κομισιόν δεν έχει σκοπό να υποβάλει πρόταση για αυτά τα θέματα. Έτσι φαίνεται. Για τις υπηρεσίε γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να προβλέψουμε καταρχήν έναν ορισμό. Ένα σαφή ορισμό, διότι γνωρίζετε πως ε, σε διάφορα κράτη-μέλη έχουν εμφανιστεί πολλά παράπονα και καλό είναι να εναρμονίσουμε τον ορισμό. Τώρα, για την κοινωνική ρήτρα και το εύρος της, θα θέλαμε να είναι λίγο πιο δεσμευτική. Αυτό βέβαια θα απαιτούσε μια περισσότερη επεξεργασία του θέματος σε βάθος. Και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα η Κομισιόν να μας, να μας είχε υποβάλει μια αρχική πρόταση. Ο Επίτροπος Μπαρνιέ έχει στόχο να διατηρήσει αυτή την, κοινωνική, την πρόταση για την κοινωνική ρήτρα. Είδατε και η έκθεση Μόντι ήταν υπέρ της ρήτας αυτής. Επίσης θα θέλαμε οι προτάσεις να είναι πιο τολμηρές σε ό,τι αφορά την νομοθεσία περί επαγγελματικής ζωής. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο μας αφορά και εμάς και τους πολίτες είναι η οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα. θα έπρεπε να αναρωτηθούμε πώς θα εφαρμοστούν τα όσα προβλέπονται. Για παράδειγμα, η επαγγελματική κάρτα. Ίσως θα ήταν πιο εύκολο ένα να καθιερώσουμε ένα σύστημα επαγγελματικών καρτών, διότι έχουμε ήδη προηγούμενα. Έχουμε για παράδειγμα τις υπηρεσιακές ταυτότητες ε, στις Βρυξέλλες. Καταλαβαίνετε ότι ε, αυτό θα μπορούσε να μην είναι τόσο δύσκολο. Ευχαριστώ. Κυρία Μωρέα και μετά ο κύριος Κρούτσμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το κείμενο έχει κάποια ε, ισχυρά σημεία στα οποία θα πρέπει να επιμείνουμε και ίσως θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και κάτι. Ε, να σας πω καταρχήν ότι το κείμενο συνδέει την ε, εξέλιξη της απασχόλησης, την αύξηση απασχόλησης με την οικονομική ανάπτυξη. Δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί η απασχόληση αν δεν εξασφαλίσουμε ανάπτυξη. Συνεπώς, κοιτάζουμε πώς θα βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω χρηματοδότησης αφενός, γιατί ε, η ανέβρεση χρηματοδότησης, ε, ανέβρεση πιστώσεων είναι δύσκολο έργο ε, και δεύτερον μέσω της, των λογιστικών αλλαγών, αλλαγών στο λογιστικό σύστημα. Η οργάνωση της εσωτερικής αγοράς όπως μας προτείνεται ε, στην οργάνωση αυτή είναι πολύ σημαντική η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας γιατί αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ την καινοτομία που είναι πολύ σημαντική ε, τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνία θα χρησιμεύσουν πολύ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ε, ζητήσουν την, να καταθέσουν αίτηση σε κάθε μία από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης για να λάβουν εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα ήταν ένα σύστημα πολύ πιο λαφρύ, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις και θα ήθελα να επανεισαχθεί το θέμα αυτό στην ε, έκθεσή μας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. χαιρετίζουμε την σημασία που δίνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, που ε, έχουν σημαντική συμβολή για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα γραφειοκρατικά εμπόδια στην Ευρώπη και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν 27 διαφορετικά γραφειοκρατικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλο ένα σημαντικό σημείο για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει που σωστά αναφέρει ο κ. Μπαλτασάρε είναι η πρόσβαση στην χρηματοδότηση. Τα, τα προγράμματα χρηματοδότηση ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να οργανώνονται χωρί γραφειοκρατικό τρόπο, ώστε να έχουν ε, εύκολη πρόσβαση σε επιχειρηματικά κεφάλαια μικρομεσαίε επιχειρήσει. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να προτείνουμε να υπάρχουν κοινωνικές ε, ρήτρες σε όλες τις συμβάσεις. Τη λέξη όλες δηλαδή θέτω κάπως σε αμφισβήτηση. Νομίζω ότι είναι καλή η πρόθεση, αλλά δεν ξέρω αν θα πρέπει ε, να πούμε όλες, σε όλες τις περιπτώσεις, γιατί αυτό δεν θα είναι εφικτό σε κάθε περίπτωση. Είναι σημαντική η συμβολή στην απασχόληση και τις κοινωνικές ε, παροχές, αλλά θα πρέπει να μιλάμε για προ εμπορικές ε, συμβάσεις, ούτως ώστε να δημιουργείται η κρίσιμη μάζα για καινοτόμα προϊόντα και να δημιουργούνται νέες αγορές και θα πρέπει ε, να έχουμε κατά νου, πούμε, ότι για θέματα κινητικότητας ε, για κάθε χώρα έχει σημασία να υπάρχουν καινοτόμα προϊόντα που θα προσφέρουν κάτι παραπάνω στην αγορά εργασίας. Ε, τέλος, για την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, στις δημόσιες συμβάσεις είναι τεράστιος ο τομέας, ένα μεγάλο πρόβλημα όπως γνωρίζουμε και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Ε, ξέρετε ότι ο ανταγωνισμός οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές, τόσο ώστε οι καταναλωτές να έχουν χαμηλότερες τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό ισχύει για τον ανταγωνισμό και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο λόγια μόνο ως δική μου συνεισφορά σε αυτή την τόσο σημαντική συζήτηση για την νέα αγορά της μικρομεσαίας επιχειρήσης και την ανάπτυξη. Η Κομισιόν ε, ανέλαβε την πρωτοβουλία να υποβάλει μέτρα για την αναζωογόνηση της νέας αγοράς και σε αυτή τη συγκυρία είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για την Small Business Act και να υπογραμμίσουμε ιδιαίτερα την ε, τροποποίηση της Small Business Act που προτείνεται να γίνει σύντομα για να δώσουμε μια πιο ισχυρή κοινωνική διάσταση στον τομέα αυτό. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν ένα τεράστιο δυναμικό της αγοράς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, για τη διατήρηση θέσεων απασχόλησης και η μεταρρύθμιση, η αναθεώρηση τη Small Business Act θα μπορούσε να αποτελέσει ένα βήμα για να διευκολύνουμε την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση για να μειώσουμε την γραφειοκρατία των μέτρων του συστήματος στο οποίο υπόκεινται και για να διευκολύνουμε τη ζωή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να μπορέσουν με μεγαλύτερη ευκολία να διατηρήσουν τις θέσεις εργασία και να δημιουργήσουν καινούριε. Μέσω αυτού του οικονομικού τομέα θα έχουμε έναν μοχλό, σοβαρό μοχλό για να ενισχύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τόσο πολύ χρειαζόμαστε στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ποιος άλλος θα ήθελε το λόγο, κύριος Κρίστοφσεν. Μπορώ να μιλήσω δανέζικα, πρόεδρε. Okay. Όχι, δεν μπορείτε να μιλήσετε δανέζικα. Αν θέλετε, μιλάτε γαλλικά. Μία ερώτηση για τον κύριο Παλτασάρε ασφαλώς είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης. Όμως ο κ. Βαλτασάρ μίλησε για ανταγωνιστικούς μισθούς. Τι εννοεί άραγε. Δεν είναι δυνατόν το εργατικό δυναμικό να το αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Γιατί υπάρχουν δικαιώματα εργασιακά δικαιώματα. Υπάρχει το δικαίωμα σε αξιοπρεπείς μισθούς, συλλογικέ συμβάσεις, ασφάλεια ε, και υγεία στο χώρο εργασίας κλπ. Συνεπώ, οι μισθοί δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται όπως αντιμετωπίζονται τα εμπορεύματα. Επίσης με ανησυχεί το πώς βλέπει η Κομισιόν τη Single Market Act. Διότι δεν λαμβάνει και πολύ υπόψη την κοινωνική ατζέντα Εμείς θα πρέπει να αντιδράσουμε. Αυτά, ευχαριστώ. Arvoisa puheenjohtaja, minä kaipaisin... Ευχαριστώ, Χρειαζόμαστε κάποιες διευκρινήσεις για το εγγράφο της Επιτροπής. Συγκεκριμένα, το σημείο 19. Ποια είναι η θέση μας. Υπάρχει μια κοινή φορολογική βάση για τις επιχειρήσεις. Μετά υπάρχει το σημείο 20 για τη στρατηγική σχετικά με το ΦΠΑ. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα. Ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάποιος αναφέρθηκε στην κοινωνική ατζέντα και ε, στη διάθεση του ΑΕΠ. Ε, ποια είναι η θέση μας επί του θέματος. Είναι λυπηρό που η Επιτροπή δεν έχει συμπεριλάβει κάτι σε σχέση με τον φόρο επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, που αποτελεί μια δυνατότητα και μάλιστα το φθινόπωρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μίλησε για το θέμα αυτό. Εκφράσαμε τη θέση μας. Στο έγγραφο αυτό, επίσης θα πρέπει να τονίσουμε ότι κάτι πρέπει να γίνει και για τους φορολογικούς παραδείσους. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Γιακονσάρη. Δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο. Ναι, συμφωνώ και εγώ με αυτήν την τελευταία πρόταση της κυρίας Γιάκων Σάρη, γιατί νομίζω ότι στο πακέτο για τα δημοσιονομικά θέματα δεν μπορούμε να καλύψουμε όλα τα σημεία, αλλά αν εμείς μπορούμε να φροντίσουμε να υπάρχει συνοχή στα όσα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα είναι χρήσιμη αυτή η συμβολή μας. στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει επιτάπητο διάφορα σημεία, μεταξύ των οποίων πολλά δεν υποστηρίζω. Όμως υπάρχει αφενός μεν η επανέναρξη της συζήτηση για την εναρμόνιση της φορολογικής ε, βάσης, για την ε, φορολογία των εταιριών, Υπάρχει μια άλλη πρόταση στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για την ε, καλύτερη ισορροπία ε, στις κεφαλαϊκές αγορές και στις αγορές εργασίας και νομίζω ότι και γι' αυτό ε, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε να μπει κάτι στο κείμενο. Πολλοί συνάδελφοι φοβούνται ότι θα χάσουμε ανταγωνιστικότητα αν έχουμε μεγαλύτερη εναρμόνιση στα φορολογικά θέματα. Αν θέλουμε όμως ε, μεγαλύτερη απασχόληση στην Ευρώπη στο μέλλον, το θέμα της ε, φορολογίας είναι κάτι που άμεσα μας ενδιαφέρει. Θα μπορούσαμε να ε, παρέμβουμε λοιπόν όχι μόνο στα θέματα της φοροδιαφυγής, που είναι μεγάλη δυσκολία για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αλλά και στο θέμα της ισορροπίας μεταξύ της φορολογίας του κεφαλαίου και της ε, φορολογίας της εργασίας. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για το σημείο 14. Όσον αφορά τα λογιστικά και αναφέρεται και η θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχει διεθνής εναρμόνιση για, τα, για τη λογιστική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θέλουμε να ελαφρύνουμε τα βάρη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και όχι να τις επιβαρύνουμε με κοινέ ε, διεθνείς διατάξεις. Για ορισμένε μικρομεσαίες επιχειρήσεις εμείς θα τίναμε να είμαστε κατά της ε, ε, ανάγκης συγκεκριμένης λογιστικής, πόσο μάλλον διεθνών λογιστικών συστημάτων. Στο σημείο 15 είναι κάτι που ανέφερε και η κυρία Γιακονσάρη. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να χρηματοδοτήσει μέσω δανείων επενδυτικά μακροπρόθεσμα σχέδια, αλλά πρέπει να υπενθυμίσουμε τα στοιχεία που υπάρχουν στην οριζόντια ρήτρα, στο άρθρο 9 της Συνθήκης της Λισαβόνας, να γίνει ένας απολογισμός ή μια προκατακτική μελέτη για το τι αναμένουμε από τέτοιες επενδύσεις όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Και για τις προτάσεις 23 και 24 σημειώνω με ικανοποίηση στο σημείο 24 το ότι λέμε το να εξασφαλίσουμε ενισχυμένη συμμετρία αυτό υπάρχει μέσα στην πρόταση της Επιτροπής. Αν δεχθούμε να συζητήσουμε τη συμμετρία αυτή, θα πρέπει αυτό να γίνει και στο θέμα των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων. Μέσω της γνωμοδότησης του κυρίου Μπαλτασάρ, λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε στην τροποποίηση της αρχικής πρότασης της Επιτροπής. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στον εισηγητή για να κλείσουμε αυτήν την πρώτη ανταλλαγή απόψεων και σας ευχαριστούμε για τις προτάσεις σας. Κύριε Παλτασάρα, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που με τις παρεμβάσεις τους εμπλουτίζουν αυτή τη συζήτηση που είναι και από δικό της ενδιαφέρουσα. Βέβαια, δεν θα είναι κάτι το καινούριο αυτό στην ενιαία αγορά αλλά σε, κατά μεγάλο μέρος ε, ε, δεν έχει πραγματοποιηθεί το σύστημα αυτό, δεν μπορεί να, εξηγεί, να εκφραστεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο πέρα από τη χώρα. Ε, αυτά τα στοιχεία που έχουμε το δείχνουν καθαρά. Μόνο ένα περιορισμένο ποσοστό επιχειρήσεων μπορεί να εργαστεί στην ενιαία αγορά να εξαγεί σε άλλες χώρες και αυτό βέβαια είναι ένα από τα όρια της αγοράς. Η νέα αγορά θα πρέπει να επιτρέπει στις επιχειρήσεις ε, έτσι γεωμετρικά να αναπτύσσονται, να ανοίγονται ε, σε νέες αγορές και να προωθούν τα προϊόντα σε όλη την Ευρώπη. Δεν γίνεται όμως δυστυχώς αυτά. Είναι απογοητευτικές αναλύσεις της Επιτροπής πάνω σε αυτό και δεν γίνεται και στην κανονική αγορά. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται στην αγορά μέσω ίντερνετ ε, και τα στοιχεία αυτά είναι απόλυτα πραγματικά. Βέβαια, μέσα σε μια χώρα οι αγορές, οι διαπραγματεύσεις μέσα του ίντερνετ είναι της τάξης του 26%. Οι επαφές αυτές είναι μόνο 7% πέρα από τα σύνορα. Δεν υπάρχει, δεν ισχύει εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει ένα μέσο που να καθησυχάζουν τον καταναλωτή για να αποκτάει προϊόντα που έρχονται από άλλη χώρα έστω και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται καθαρά ότι στην κατάσταση αυτή οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι πολυεθνικές, εκείνες μπορούν να είναι παρούσες γύρω-γύρω ε, παντού, διεθνώς ε, μεγάλες ιταλικές, γερμανικές, γαλλικές. Μόνο οι μεγάλες, οι μικρές δεν τα καταφέρνουν. Έστω και αν η ποιότητα των προϊόντων είναι άριστη, αλλά η ενιαία αγορά εκεί δεν έχουν πρόσβαση οι μικρές επιχειρήσεις. Και είναι από τα σημεία τα οποία συζητούνται από τα θέματα που μας απασχολούν και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κατευθύνουμε τις προσπάθειες μας ακριβώς ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να εργάζονται και εκεί. Τα δικαιώματα των καταναλωτών επίσης. Αυτά θα εξεταστούν στην Νομική Επιτροπή σε λίγες μέρες και θα είναι ένα νομικό ε, σύνολο που θα βοηθήσει και τις προοπτικές επιτροπής ε, να παρέμβει για να υπάρξει ένας οργανισμός, ε, ένα παρατηρητήριο ώστε να διευκολυνθούν οι επαφές και οι αγορές μέσω ίντερνετ θα είναι και μια άλλη λύση επίσης. Να βρεθούν λοιπόν μέσα για να διευκολύνουν την επαφή μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτών και ακριβώς επιχειρήσεις μέσα σε μια ενιαία αγορά με τρομέρες δυνατότητες που δεν αξιοποιούνται όμως, δεν χρησιμοποιούνται. Και το θέμα της ε, ε, ε αποκλειστικής ακριβώς και αυτό δεν έχει προχωρήσει. Υπάρχει μια ενισχυμένη συνεργασία και βέβαια μόνο για τα επίσημα αυτά στοιχεία θα ψηφιστεί στην νομική επιτροπή σε δύο μέρες μέσα και ε, ξέρουμε πως έχει όλη πορεία ε, τι θα γίνει με την ενισχυμένη συνεργασία και τι θα γίνει με αυτά που θα πει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά και χρήσιμα στο σύστημα των επιχειρήσεών μας και αποτελεί βέβαια και κάτι ε, που θα μπορούσε να πετύχει η Επιτροπή τη χρονιά αυτή. Έχουμε και άλλες πτυχές, ε, κυρίως όσον αφορά τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, ε, κοινού ενδιαφέροντος, την πρόταση την 25, που κατά κάποιο τρόπο έχει αναλυφθεί η υποχρέωση να συντάξει μια ανακοίνωση και να προωθηθούν ε, ενέργειες οι οποίες κατά κάποιο τρόπο θα χρησιμεύσουν για να ε, λυθεί αυτός ο γόρδιος δεσμός, ε, ε, αυτά που η πρόσφατη οδηγία δεν κατάφερε να επιλύσει. Πολλές πτυχές λοιπόν στο κείμενο της Επιτροπής ε, που χρειάζεται να προωθηθούν, να συμπληρωθούν, να πραγματοποιηθούν και αναφορές για το φορολογικό σύστημα. Εγώ συνεχίζομαι να υπερασπίζομαι δική μου η άποψη εδώ με ένα ενιονόμισμα σε αυτή την ένωση ε, στα συστήματα και τα φορολογικά δεν θα πρέπει να διαφέρουν τόσο πολύ το ένα από το άλλο. Να μην έχουμε 27 κράτη-μέλη που να έχουμε συνταξιοδοτικό και φορολογικό σύστημα εντελώς διαφορετικό. Γιατί πολλές φορές αυτές οι κρίσεις, ε, η, ε, το αίτιο είναι ακριβώς την αδυναμία ενός κράτους μέλους που δεν καταφέρνει να πετύχει αυτούς τους στόχους για ας πούμε σε ποια ηλικία ε, συνταξιοδότηση ε, και συμβαίνει και με το μέσο όρο στην Ευρώπη και για το φορολογικό σύστημα. Υπάρχει μια φοροδιαφυγική ιδιαίτερα υψηλή και τα κράτη-μέλη φαίνεται ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μετά το δημόσιο χρέος και να έχουν πόρους μέσα σε ένα σύστημα που να είναι δικαιότερο. Συνολικά, κατά την άποψή μου, εντάξει θα μπορούσε κανείς να δει πώς θα βοηθήσει για να βελτιώσει ακόμα περισσότερο το κείμενο αυτό και με αναφόρες που να μην έχουν άμεση ιδιαίτερη σχέση με το σύστημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στην τελευταία παράγραφο, ας πούμε, για να ολοκληρώσω για, μετά από την υπόδειξη της ε, Προέδρου στην τελευταία παράγραφο της ε, έκθεσης ε, συμπεριλάβα μια σύντομη αναφορά σε αυτή την ανάγκη ότι οι διεθνείς συμφωνίες που κλείνονται εκεί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη συμμετρία κοινωνικής φύσεως, δηλαδή ότι ισχύει αυτή η ανάγκη από δικής μας πλευράς να ευνοήσουμε μια ανάπτυξη κοινωνικής φύσεως ε, που να αξιοποιεί και να βοηθάει τους εργαζόμενους και στα δικαιώματά τους και όταν ε, διαπραγματευόμαστε με άλλα κράτη. Εντάξει, στην Ευρώπη υπάρχει μια κάποια εγγύηση κοινωνικής προστασίας κλπ. Και, και με, διαπραγματευόμαστε με άλλες χώρες που υπάρχουν εντελώ διαφορετικά συστήματα προστασίας των εργαζομένων ή δεν υπάρχουν καθόλου. Και ακόμα για τον δανό συνάδελφο ανταγωνιστική μισθή δεν σημαίνει χαμηλή μισθή για να παραμείνει κανείς ε, όπως πρέπει στην αγορά, μειώνοντας το κόστος ε, για να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια κάποιου στελέχους ε, από τη Fiat στο Τωρίνο. Να είναι κάποιος έτσι πάτερ φαμίλιας, να μπορεί να εγγυηθεί ένα κάποιο εισόδημα σε ένα εργαζόμενο και που στο τέλος ε, της δουλειάς του να βλέπει τον καρπό της εργασίας του. Άρα λοιπόν να βοηθιέται και ο καταναλωτής. Ε, να μην έχουμε μόνο μια προσοχή που να αποδίδουμε στα πλαίσια του συστήματος. Και ακόμα ε, μέχρι τις 6 αύριο 26 Ιανουαρίου η προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Ναι, το μεσημέρι, το μεσημέρι διορθώνει ο Σας ευχαριστώ. Ναι. Για τους καταναλωτές, οι καταναλωτές συχνά είναι και μισθωτοί βέβαια. Σε ευχαριστούμε πάντως ε, και που μας υπενθυμίσατε την ημερομηνία υποβολής τροπολογιών. 26 Ιανουαρίου είχε οριστεί τελικά στις 6 το αργά το απόγευμα. Έχουμε πολλή δουλειά και στο όλο χρονοδιάγραμμά μας, αλλά η Επιτροπή μας θέλει να σεβαστεί αυτό το χρονοδιάγραμμα, ώστε το Μάρτιο να καταλήξουμε στην Ολομέλεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό που επιθυμεί είναι να προχωρήσει τάχιστα στο σύνολο αυτών και θα ήθελε επίσης να ξέρει ποια είναι η απόψή μας πάνω σε αυτό. Και 26 Ιανουαρίου αύριο μέχρι τις 6 αυτές ε, και 1η Φεβρουαρίου θα το εξετάσουμε και 14 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο, ίσως ως συνάδελφοι δεν τους αρέσει, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα με το ρυθμό των υποχρεωτικών των εργασιών μας των κοινοβουλευτικών και στη συνέχεια θα έχουμε 14 μέρες για να χτενίσουμε κάπως το θέμα και να δούμε πώς η Ερμόδια Επιτροπή θα λάβει υπόψη της ε, την γνωμοδότηση τη δική μας. Πάμε τώρα στο δεύτερο σημείο του όλου συνόλου, του όλου πακέτου. Ο κ. Κρόιτσμαν είναι ο εισηγητής, έχει να κάνει με την εταιρική σχέση, την εσωτερική αγορά και για το θέμα αυτό θα έπρεπε κανονικά να έχουμε μια ενισχυμένη συνεργασία, δηλαδή μια επιτροπή που θα συνεργάζεται μαζί μας και η Επιτροπή ΙΝΚΟ ακριβώς θα πρέπει να λάβει υπόψη διάφορες ε, απόψεις διαφόρων επιτροπών πάνω σε αυτό. Καμία Τέλος πάντων, άτυπα, άτυπα να γνωρίζετε ότι θα είναι κάτι το καινοτόμο, ε, θα είμαστε συνεργαζόμενοι επιτροπή έτσι άτυπα και θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα πράγματα για την έκθεση του κύριου Κρόιτσμαν. Ε, έχει τον λόγο ο κύριος Κρόιτσμαν για να μας κάνει την εισηγήθησή του. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Στη γνωμοδότησή μου τονίζω την ανάγκη για τον ανταγωνισμό στην ε, ενιαία αγορά. Αυτό είναι κάτι που θα υλοποιηθεί όταν ε, κατορθώσει να δώσει και στους πολίτες και στις επιχειρήσεις γενικά, συμπεριλαμβανομένων και των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την αίσθηση ότι στην καθημερινότητα προσφέρει πλεονεκτήματα. Αυτό οφείλεται, θα οφείλεται και στη σωστή διακυβέρνηση που είναι απαραίτητη για την επίταξη των οικονομικών και κοινωνικών στόχων της ενιαίας αγοράς. Εδώ συμπεριλαμβάνεται όσον αφορά την Επιτροπή Απασχόλησης. Ε, ε, εδώ συμπεριλαμβάνεται και η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, υψηλό επίπεδο απασχόληση, κατάλληλη κοινωνική προστασία, καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης, γιατί αυτά αποτελούν τη βάση των δυνατοτήτων ε, απασχόλησης και παράλληλα αποτελούν και τη βάση για την απασχόληση ε, και για τη δημιουργία μεγαλύτερη απασχόληση στην Ευρώπη. Επίση, τονίζω το σημαντικό ρόλο των δικτύων υποστήριξη όπω είναι το ΕΡΕΣ και το Solvit για τη σωστή λειτουργία τη ενιαία αγορά ε, όταν οι πολίτε ε, θα προσπαθούν να ζητήσουν θέσεις απασχόληση σε άλλε χώρε και θα θέλουν να λύσουν τα προβλήματά του με τι δημόσιε αρχέ. Και για την απασχόληση θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία το να υπάρχουν εργαζόμενοι μέσα στην Ευρώπη με μεγαλύτερη ευελιξία. Ξέρω ότι δεν είναι απλό, ξέρω ότι εξαρτάται από τα διαφορετικά κοινωνικά και πολιτιστικά συστήματα, ε, είναι διαφορετική φιλοσοφία, διαφορετική γλώσσα και υπάρχουν ε, και γλωσσικοί φραγμοί, αλλά είναι πολύ σημαντικό να παρέχεται η δυνατότητα για να παρέχονται ευκαιρίες από το άνοιγμα και προς τις χώρες τη Ανατολικής Ευρώπης για να υπάρξει απασχόληση στις χώρες όπου υπάρχει ζήτηση. Σκέφτομαι, α πούμε, τη Γερμανία σαν παράδειγμα. Υπάρχουν ε, χιλιάδες ε, ε, θέσεις απασχόλησης για εξειδικευμένους ε, και σε άλλες χώρες υπάρχουν προβλήματα απασχόλησης. Υπάρχει λοιπόν η λύση της ευελιξίας που θα επιφέρει μια ισορροπία μεταξύ της αναζήτησης θέσεων απασχόλησης και της προσφοράς θέσεων είναι ε, σημαντικό να συμμετέχουν ε, όλοι οι ενδιαφερόμενοι στο ε, σχεδιασμό και την εφαρμογή των μέτρων χωρίς γραφειοκρατία. Δεν θέλουμε να υπάρχει ευρωσκεπτικισμός. Όταν βλέπουν οι άνθρωποι ότι αυτό το οποίο κάνουμε εδώ στην Ευρώπη τους προσφέρει ένα πλεονέκτημα στην καθημερινή του ζωή, όταν βλέπουν την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα υπάρξει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, καλούμε την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τους κοινωνικούς εταίρους, ιδιαίτερα κατά την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας και να υποστηρίξει την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας στους τομείς αυτούς τονίζω για άλλη μια φορά τη σημασία που έχει η εταιρική σχέση με τους ε, κοινωνικούς εταίρους. Είναι πολύ καλή εμπειρία που έχουμε στη Γερμανία και πάντοτε με τους κοινωνικούς εταίρους επιτυγχάνουμε, με τα συνδικάτα κατέστη μόνο δυνατόν να συμφωνήσουμε, παραδείγματο χάρη διατάξει ε, για το περιορισμένο χρόνο εργασία, κάτι το οποίο ε, βοήθησε στη Γερμανία τη δημιουργία θέσεων απασχόληση και ήταν ε, μια δράση πρότυπο που μόνο χάρη στην εταιρική σχέση με του κοινωνικού εταίρου μπορέσαμε να το επιτύχουμε. Νομίζω ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη λοιπόν θα είναι πολύ σημαντικό και οι επιχειρήσει και οι εργαζόμενοι να συνεργαστούν προ την ίδια κατεύθυνση για να επιτύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κάποιος που θα ήθελε να παρέμβει, να έχετε το λόγο. Η κυρία Γιακονσόρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ νομίζω ότι υπάρχει καλή βάση για τη γνωμοδότησή μας. Επιμένουμε για το ρόλο των κοινωνικών εταίρων και για τη σημασία της κοινωνικής διάστασης. Μιλάμε για την ανταγωνιστικότητα και για την κοινωνική οικονομία της αγοράς. Ιδιαίτερα σημαντικό σημείο. Όπως είπε ο εισηγητής, υπάρχει το δίκτυο Solvit, το οποίο είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι γνωστό από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι πολύ λίγο γνωστό το δίκτυο Solvit. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να λάβουμε μέτρα, ούτως ώστε το δίκτυο αυτό να γίνει ευρύτερα γνωστό. Και η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη πρέπει εδώ να παίξουν κάποιο ρόλο. Πάντως είναι καλή βάση για περαιτέρω εργασία αυτή η πρόταση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που άκουσα αυτές τις παρεμβάσεις ε, γιατί το κείμενο Κρότσμαν ε, αποτελεί άριστη βάση εργασίας Η Ευρώπη είναι τη προς τιμή της που σε αυτές τις ε, ώρες κρίσης ε, στην ενιαία αγορά την ευρωπαϊκή βλέπουμε έτσι ότι έχουμε αυτή την κοινωνική πτυχή που συνδέεται αναπόσπαστα με την οικονομική πτυχή. Και μέσω του λογοκειμένου η κοινωνική οικονομία της αγοράς λαμβάνει το νόημά της και από το 1992 έτσι μπορούμε να έχουμε ένα νέο κείμενο μετά τώρα εδώ. Ευχαριστώ κύριε Κρόιτσμαν. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το ποσοστό το υψηλό απασχόλησης να διατηρηθεί και ακόμα οι μεταρρυθμίσεις αυτές να γίνουν σε απόλυτη με με τους κοινωνικούς εταίρους και να ενισχυθεί και ο κοινωνικός διάλογος της επιχειρήσης και ακόμα ένα τελευταίο σημείο εδώ η εμπιστοσύνη σε αυτή την αγορά περνάει, να μην ξεχνάμε, μέσω μιας καλής επικοινωνίας με το κοινό και με τους κατανοτές και με τις επιχειρήσεις. Μια καλή πληροφορία ότι είναι καλά βασισμένη αυτή η νέα αγορά και έτσι διατηρείται εμπιστοσύνη στην αγορά σε αυτή την παγκοσμιοποίηση. Ε, στο χαρακτήρα αυτό το καινούργιο που μπορούν να τα κακοποιήσουν. Ευχαριστούμε κύριε Κρόιτσμαν που θίξατε αυτά σε μια κλειδιά ε, στην αυτή την ενιαία αγορά και στο πώς ε, τοποθετείτε το θέμα. Oui. Merci. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Εδώ. Νομίζω ότι με αυτό το πακέτο της Single Market Act εκφράζουμε την βούληση αλλά έχουμε και την ευκαιρία να ξανα εξασφαλίσουμε την ισορροπία της εσωτερικής ε, αγοράς. Η έκθεση Μόντι επιβεβαιώνει ότι η αγορά αυτή δεν βρίσκεται σε ισορροπία ε, εις βάρος των πολιτών και της κοινωνικής πτυχής της. Συνεπώς, πέραν των τριών κεφαλαίων που έχουμε καθορίσει προκειμένου να διευκολύνουμε τις συζητήσεις και θα τα συζητήσουμε το ένα κατόπιν το άλλο διαδοχικά. Χρειάζεται να υιοθετήσουμε και μια οριζόντια προσέγγιση των τριών κεφαλαίων. Δηλαδή, πρόοδος και απλοποίησης υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα πρέπει να εξισορροπείται από πρόοδο στο κοινωνικό τομέα. Σύγκληση των λογιστικών προτύπων, δηλαδή ε, διασύνδεση των μεμπορικών μητρών και λοιπά αφενός, αλλά από την άλλη μεριά και ταυτόχρονα θα πρέπει μέσω της αναθεώρησης της ε, ε, οδηγίας για τις αποσπάσεις να εξασφαλίσουμε τη σύγκληση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Για παράδειγμα, επιχειρήσεις, ε, ε Ευρωπαϊκές Επιτροπές Επιχειρήσεων, ανακλάδο οι, οι βιομηχανικές... Ε, ε, ε, οι εργασιακές αλλαγές θα πρέπει να υπόκεινται στην εξέταση των ε, επιτροπών ε, επιχειρήσεων κλπ. Χρειάζεται λοιπόν μια οριζόντια προσέγγιση, διότι αν δούμε κατακαιρματισμένες προτάσεις μία προς μία και διαδοχικά, υπάρχει περίπτωση να καταλήξουμε ξανά σε κάτι που να μην είναι ισορροπημένο. Γιατί η κοινωνική πρόοδος, η πρόοδος στα κοινωνικά δικαιώματα δεν θα πρέπει να είναι απλώς πράσινες βίβλοι και λόγια, κούφια. Θα πρέπει η απλοποίηση να πηγαίνει χέρι-χέρι με την ε, προγωγή των κοινωνικών δικαιωμάτων. Αυτό που να το πούμε από τώρα, έτσι ώστε η Κομισιό να ξέρει ότι αυτά δύο θα πρέπει να τα δει μαζί. Για την ενέργεια, για παράδειγμα, υπάρχουν προτάσεις για φορολόγηση της ενέργειας, ένα πρόγραμμα ενεργειακής αποδοτικότητας. Θα πρέπει όμως ταυτόχρονα να δούμε προτάσεις όχι μόνο για τις υποδομές, τις ενεργειακές υποδομές, αλλά και για το πώς θα λειτουργεί αυτή η εσωτερική αγορά ενέργειας. Αυτή η εσωτερική αγορά ενέργειας, η ενιαία αγορά ενέργειας, θα πρέπει να συμπληρωθεί με προτάσεις εγγύησης, εγγύησεων, κοινωνικών εγγύησεων. Ε, μια ενεργειακή ασπίδα, ξέρω εσείς πρόεδρε, είναι το θέμα αυτό ε, πολύ ε, ε, δικό σας ε, επίσης ε, να μιλήσουμε για τις ε, κρατικές επενδύσεις το τομέα ενέργειας κλπ. Μετά η πρόταση 9 για, για μια επιτροπή ψηλού επίπεδου σε, σε για, την για τη βοήθεια των επιχειρήσεων νομίζω ότι θα πρέπει μια παρόμοια επιτροπή να δημιουργηθεί και για την κοινωνική πτυχή, έτσι ώστε να προχωράμε παράλληλα. Σε ό,τι αφορά τις, ε, ε, ε κοινωνικές ε, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, ε, νομίζω ότι και εδώ έχουμε πολλές προτάσεις να κάνουμε. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα δράσης. Το Κοινοβούλιο μπορεί να υποβάλει τις προτάσεις για να δούμε προς τα πού θα κινηθούν προς τα πού θα κινηθούμε το, στο μέλλον. Για τη διακυβέρνηση, εντάξει θα μιλήσουμε λίγο αργότερα, αλλά... δεν είμαστε σε αυτό το θέμα, καλά. Εγώ θα ήθελα να ε, προτείνω Επιτροπή Υψηλού Επίπεδου για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής ωφέλειας, Επιτροπές Επιχειρήσεων, Ευρωπαϊκές Επιτροπές Επιχειρήσεων, ε, διατάξεις έτσι ώστε ο τομεακός, ο κλαδικός ε, διάλογος για τις επενδύσεις, για τις και κλπ. να είναι αποτελεσματικός και επιτροπές ελέγχου για μια ενεργειακή ασπίδα και την Ευρωπαϊκή Χάρτα Μεταφορών. Ευχαριστώ. Euh, Θέλει κανείς άλλο το λόγο για το κομμάτι διακυβέρνησης του πακέτου. Αν όχι, να κάνω εγώ κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Κρόιτσμαν για την ε, παρουσίασή του. Στην πρόταση Κομισιόν υπάρχουν νομίζω πολλά θετικά για μας. Ταυτόχρονα όμως, αν δεν μου ξέχει κάτι, δεν βλέπω ότι, την ιδέα ότι για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ε, θα πρέπει η νομοθεσία να σέβεται την ποικιλία των ε, διαφόρων νομικών καθεστώτων που επικρατούν. Δηλαδή, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τον ιστό της οικονομικής, της κοινωνικής οικονομίας ε, των χώρων κρατών μελών μας και αυτός ο ιστός θα πρέπει να είναι συμβατός με τα νομοθετήματα που προτείνει η Κομισιόν. Νομίζω ότι αυτό είναι ανησυχία και της Επιτροπής μας για τα θέματα απασχόλησης. Για την πρόταση 47 για το σεβασμό των κανόνων της εσωτερικής αγοράς Νομίζω ότι συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό από την άλλη μεριά, όταν συζητούσαμε την συμφωνία πλαίσιο στην αρχή της θητείας μας, είχαμε δει, είχαμε συζητήσει το πώς η Κομισιόν θα προσφεύγει στο δικαστήριο για αθέτηση των κανόνων της, ε, ε των ευρωπαϊκών κανόνων, ιδιαίτερα για κοινωνικά ζητήματα ε, ή πώς θα ξεκινάει η διαδικασία σε παραβάση για τέτοια θέματα. Θα πρέπει να το επαναλάβουμε εδώ γιατί βλέποντας τις ε, προσφυγές ε, της ε, Κομισιόν, η παράβαση κοινωνικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας είναι πολύ σπάνια ως αίτιο. Για την πρόταση 48 επιμένεται για την διάσταση κοινωνικού διαλόγου, κύριε Σίγητα. Αυτό που μου είναι όμως εντυπωσιακό είναι ότι ο διάλογος με την κοινωνία των πολιτών είναι πάνω-πάνω, είναι πρώτος-πρώτος. Συμφωνώ, συμφωνώ με το διάλογο με την κοινωνία των πολιτών. Συμφωνώ να συμπεριληφθούν και οι μη κυβερνητικέ οργανώσει σε αυτόν τον κατάλογο και να λαμβάνουν την υπόψη και οι ε, περιφερειακές οργανώσεις. Όμως, το θέμα του κοινωνικού διαλόγου είναι το πιο σημαντικό. Και για να έχουμε, πολύ να έχουμε σωστή ισορροπία και καλή ιεραρχία χρειάζεται να είναι πρώτο πρώτος ο κοινωνικός διάλογο. Γιατί αυτή τη στιγμή λέμε πρώτα οι καταναλωτέ, μετά οι μη κυβερνητικέ οργανώσει και στο τέλο βάζετε το, τα συνδικάτα. Νομίζω αντίστροφα θα πρέπει να αναφερθούν. Αυτή ήταν η δική μου άποψη. τις προτάσεις της κυρίας Καστέξη θα τις δούμε όταν συζητήσουμε την τρίτη γνωμοδότηση. Κύριε Κρούτ, ε, ε, Κρέουτσμαν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις πολύ επικοδομητικές παρεμβάσεις τους. Νομίζω ότι δείχνουν ότι βρισκόμαστε στη σωστή οδό. Συμφωνώ με αυτό που είπατε για το Solvit, ότι το Solvit ε, είναι πολύ λίγο γνωστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς, στην οποία είμαι μέλος, προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ε, ενημέρωση των πολιτών στα κράτη-μέλη για τη διαθεσιμότητα του Solvit, γιατί το Solvit είναι ένα καλό μέσο και σε κάποια κράτη-μέλη λειτουργεί το Solvit, σε άλλα κράτη-μέλη υπάρχουν πολλές ελλείψεις και έχετε δίκιο Πρέπει να βελτιώσουμε την επίγνωση των πολιτών και να το χρησιμοποιούν περισσότερο. Ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου. Συμφωνώ με αυτό που είπατε, Πρόεδρε. Από την πλευρά της προστασίας των καταναλωτών και της εσωτερικής αγοράς, που εγώ, το βλέπουμε διαφορετικά από ότι ε, στην Επιτροπή Απασχόλησης και θα πρέπει το κοινωνικό διάλογο να το βάλουμε στο επίκεντρο. Ε, Υπάρχει στη Γερμανία η δυνατότητα της ε, συναπόφασης, της συμμετοχής των ε, εργαζομένων και πρέπει ε, να, να δούμε πού υπάρχει η προθυμία να δημιουργείται κοινωνικός διάλογος και συμμετοχή των εργαζομένων. Είναι διαφορετικές οι δομές σε κάθε χώρα. Εδώ, ήδη από τη συνθήκη της Λισαβόνας υπάρχουν κάποιες, κάποιοι περιορισμοί. Τα κοινωνικά θέματα είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. και νομίζω ότι ε, αυτό ε, μπορεί να αποτελέσει έλλειψη για τα κράτη-μέλη, γιατί αυτό που θα έπρεπε να είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών μας είναι να εντείνουμε τον κοινωνικό διάλογο υπάρχουν, ε, υπάρχει ανισορροπία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ αναφέρω συνεχώς τη Γερμανία, αλλά ξέρω ότι από την πλευρά της Γερμανίας αυτό δίνει τη δυνατότητα ε, στο να έχουμε συμμετοχή των εργαζομένων ε, και ισομερή λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο αυτής της εταιρική σχέσης. Χωρίς ε, την κοινωνική εταιρική σχέση δεν θα μπορούσαμε να έχουμε την κοινωνική ειρήνη που έχουμε στη Γερμανία. Αυτό το τονίζω για άλλη μια φορά. Θα είχαμε ε, πολύ χειρότερες συνθήκες και νομίζω ότι ο κοινωνικός διάλογος είναι αυτό που παίζει τον καθοριστικό ρόλο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ε, σωστή οικονομία και στην κοινωνική ειρήνη. Η συμμετοχή των εργαζομένων είναι αυτή η οποία έχει βοηθήσει στην πρόθεση των συμφερόντων όλων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ο ίδιος λόγος, η ίδια τιμωρία. Ακριβώς ε, ακολουθούμε την άποψή σας και το ίδιο χρονοδιάγραμμα όπως και για τον κύριο Μπαλτάσαρ. 26 ε, Ιανουαρίου στις 6 προθεσμία υποβολή τροπολογιών. Πάμε τώρα το τρίτο μέρος αυτής της δέσμης. Η κυρία Γιακονσάρη έχει το λόγο για την αγορά για τους Ευρωπαίους και ακούστε κυρία μου εκεί ε, θα έχουμε να κάνουμε με τις ε, υπηρεσίες ε, κοινοφιλούς ενδιαφέροντες. Έχει το λόγο. Ναι. Ακούστε. Αρχίζω να μαθαίνω γαλλικά και παρακολούθησα όσα υπόθηκα πριν από λίγο που, έχει σχέση, που έχουν σχέση με το σημείο αυτό, με την ενιαία αυτή αγορά και με τους πολίτες. Είναι πολύ σημαντικό σημείο, όπως είπα και προηγουμένως, και καλό θα ήταν αυτή η έννοια να διευρυνθεί για την αιτία αγορά και οι πολίτες να καταλάβουν ότι αυτό αφορά και την προστασία των κάτων και την ε, μετακίνηση, την κινητικότητα, όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τους πολίτες. νέα αγορά για τους ε, πολίτες λοιπόν. Πρόκειται για ένα τρομερά σημαντικό θέμα. Λόγω της σημασίας του ακριβώς ε, να σας πω ότι σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εμείς ε, εδώ δεν έχουμε και αρκετές προτάσεις νομοθετικές μέχρι τώρα και αναφέρομαι στις υπηρεσίες οικονομικού γενικού ενδιαφέροντος. Το επαναλαμβάνω πάντως ότι είμαι απογοητευμένοι μετά από διάφορες υποσχέσεις για επαφή, επικοινωνία, διάφορα στο λοφάσμα, αλλά όχι ενδείξεις όσον αφορά μια νομοθετικής φύσεως πρόταση. Τίποτα. Και άλλο ένα στοιχείο που με κάνει να απογοητεύομαι. Οι κοινωνικές υπηρεσίες, έτσι, παρόμοιο γενικό ενδιαφέροντος, Όλα αυτά επιφανειακά αντιμετωπίζονται σε αυτό το έγγραφο της Επιτροπής. Ίσως θα πρέπει κάπως καλύτερα να τα προσδιορίσουμε αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πριν από λίγο μίλησα για την ρήτρα την κοινωνική. Μίλησα για τον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ίσως για τα δύο αυτά σημεία χρειάζεται να συμφωνήσουμε ώστε να έχουμε μια κοινωνική δεσμευτική ρήτρα. Σε κάθε σημείο νομοθετικό και όλα αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν αντί να αρκείται κανείς εντάξει σε λεπτομεριακές αναλύσεις ε, των επιπτώσεων λοιπά, όλων αυτών που έχουν ισχύσει, όπως μας προτείνει η Επιτροπή. Πρόκειται, κατά την άποψή μας, για ένα σημαντικό σημείο. Τώρα, στο έγγραφο αυτό για τις συντάξεις. Μιλάμε για εθνικής φύσεως αρμοδιότητα. Ναι. Διαφέρει ιδιαίτερα η κατάσταση από τη μία χώρα στην άλλη, ανάλογα ακριβώς με το σύστημα συνταξιοδότησης. Πάντως θα πρέπει να επιμείνουμε ιδιαίτερα όσον αφορά τη διάρκεια αυτού του συστήματος συνταξιοδότησης. Η δική μου η πολιτική ομάδα είναι υπέρ του το συνταξιοδοτικό αυτό σύστημα να αποτελέσει μέρας του πρώτου πυλώνα. Δεν θα πρέπει όλα αυτά να τα κρύβουμε κάτω από το χαλάκι. Για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε καλά, αυτό να λειτουργήσει καλά στα πλαίσια του πρώτου πυλώνα, χρειάζεται να αποτελέσει και προτεραιότητα. Πριν από λίγο, επίσης, επέμεινα σε κάτι. Έλεγε ο τίτλος «Ενιαία αγορά για τον Ευρωπαίο πολίτη». Καλό, αλλά στα πλαίσια αυτά οτιδήποτε έχει να κάνει με τα επαγγελματικά προσόντα και την αναγνώρισή τους, αυτό είναι ζωτική σημασία. Εντάξει, εδώ πρέπει να δούμε αυτές τις έννοιες και περιμένουμε για την επόμενη χρονιά μια πρόταση οδηγίας. Αλλά νομίζω ότι θα αποτελέσει δοκιμή ιδιαίτερα σημαντική, κυρίως για το πώς θα το πάρουν αυτό ε, οι Ευρωπαίοι πολίτες. Στα πλαίσια αυτό αναφέρεται αυτή η αυτό το επαγγελματικό δελτίο. Το μέσο αυτό όμως να βοηθήσουμε να είναι απλό και αποτελεσματικό, γιατί με αυτό το μέσο θα μπορέσουμε σε να αντιπαλέψουμε την ε, παράνομη εργασία και ξέρουμε ότι στις οικοδομές στην Ευρώπη το 20% είναι από παράνομο εργαζόμενος εκεί. Αυτά είναι ορισμένα από τα στοιχεία που θα ήθελα να προσθέσω σε όσα είπα προηγουμένως ε, και ίσως ε, δεν ε, τα είπα όλα αυτά που έπρεπε σε αυτά λίγο προηγουμένως. Πάντως θεωρώ, α και κάτι άλλο, νομίζω ότι και 26 Ιανουαρίου ισχύει για την υποβολή τροπολογιών στα προθεσμία, έτσι. Κάποιος θα επιθυμούσε το λόγο, ρωτάει. Καστέξ, Θέλετε να πείτε κάτι. Όχι, δεν χρειάζεται αυτό να το επαναλάβω, έτσι. Νομίζω ότι όλοι οι συναδελφοί θα έχουν κάνει την επιλογή τους και τις προτάσεις μου θα τις έχουν βάλει στο σωστό, το, τη σωστή τη θηρίδα. Κύριε κύριος Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με το σχέδιο γνωμοδότησης γιατί υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες. Ε, φιλελεύθεροι. δεν θέλουν να είναι αντιπαραγωγικοί για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αλλά ε, για τα θέματα των ε, ε, υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος υπάρχουν πολλά θέματα γιατί σε διάφορες χώρες είναι διαφορετικά οργανωμένες αυτές οι υπηρεσίε. και πρέπει να προσέξουμε σε αυτόν τον τομέα επακριβώ ε, να προσέξουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές ε, δομές. Δεν θέλουμε να έχουμε ε, ενοποίηση και εναρμόνιση σε χαμηλότερο επίπεδο, όταν υπάρχει υψηλή προστασία των εργαζομένων σε κάποιο κράτος μέλος, να μην υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφεί αυτή η υψηλότερη προστασία χάρη της ομοιομορφίας. Ο στόχος μας πρέπει να είναι εκεί όπου υπάρχουν ε, θετικά ε, σημεία να τα διατηρήσουμε και εκεί όπου υπάρχουν μειονεκτήματα για τους εργαζομένους να τα, να τα αντιμετωπίσουμε. θα πρέπει να είναι πάντως υψηλής ποιότητας ε, και να υπάρχει πρόσβαση προς όλους. Και το εργαλείο, το toolbox που, που προτείνεται από την Επιτροπή για την χρηματοδότηση, για τις δημόσιες συμβάσεις ε, κλπ. είναι θέμα το οποίο το βρίσκω θετικό η ανάπτυξη υποδομών μεγάλων δικτύων στον τομέα της ενέργειας και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει μεγάλη σημασία σε αυτό το τομέα. Και η πρόταση της Επιτροπής για το θέμα των συχνοτήτων και ε, η χρήση του φάσματος 800 MHz ε, είναι πολύ σημαντική. στο μέλλον αυτά θα είναι θέματα τα οποία θα είναι προφανή όπως σήμερα για μας είναι το να έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα και τρέχουμε νερό στα σπίτια μας. Το να έχουμε γρήγορο ευρυζωνικό διαδίκτυο σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και θα υπάρχουν πολλές δυνατότητες κατά αυτόν τον τρόπο και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τους απασχολούμενους. Ε, δεν θα χρειάζεται να βρίσκονται όλοι σε μεγάλα αστικά κέντρα. Θα μπορεί κανείς να ε, ζει και να εργάζεται σε περιοχέ τη ε, υπαίθρου υποφελούμενο από το ψηφιακό μέρισμα. Η οριζόντια κοινωνική ρήτρα είναι ένα άλλο σημείο που πρέπει να προσέξουμε. Και θα πρέπει να προσέξουμε τις κοινωνικές επιπτώσεις. Χαιρετίζουμε την πρόταση της Επιτροπής, αλλά θα πρέπει να δούμε ακριβώς ε, τι γίνεται με την κοινωνική ρήτρα. Και Όσον αφορά το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, είναι πολλά τα θέματα που αντιμετωπίζει το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Πολύ συχνά υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση και γι' αυτό ζητάμε να υπάρχει ένα ειδικό κοινωνικό τμήμα του δικαστηρίου που να ασχολείται με το εργατικό και το κοινωνικό δίκαιο. επανέρχομαι επίσης στο θέμα της εταιρική σχέσης με τους κοινωνικούς εταίρους. Οι κοινωνικοί εταίροι ξέρουν τι είναι καλό για τους εργαζομένους στις επιχειρήσεις, γνωρίζουν τα προβλήματα και μπορούν να τα λύσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και θα κάναμε μεγάλο λάθος εάν όλα αυτά τα ζητήματα προσπαθήσουμε εμείς να τα ρυθμίσουμε μακριά από τους κοινωνικούς εταίρους, κάπου απομονωμένα στην Ευρώπη. Εκεί όπου υπάρχουν οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να τους αξιοποιήσουμε. Η κινητικότητα είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο επίσης για την ενιαία αγορά. Ε, και στις ε, περιοχές ε, όπου υπάρχουν διασυνοριακές υπηρεσίες νομίζω ότι οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από τη συνεργασία. Χρειάζεται και κατάλληλη ενημέρωση των επιχειρήσεων και των κοινωνικών εταίρων και επίσης η κοινωνική ευθύνη είναι κάτι το οποίο τονίζει η Επιτροπή και τονίζουμε και εμείς και θα πρέπει η Επιτροπή να προτείνει νέες δεσμευτικές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις και ο στόχος εδώ θα έπρεπε ε, να, να είναι και η ισότιμη συμμετοχή όλων και μεγαλύτερη συμμετοχή και των γυναικών ε, δεν θέλουμε να έχουμε δεσμευτικά Δεσμευτικέ ποσοστώσει για τη συμμετοχή των γυναικών σε διοικητικά συμβούλια, παραδείγματο χάρη, αλλά νομίζω ότι μπορεί ε, να ρυθμιστεί με μη δεσμευτικέ διατάξεις, ε, ασκώντα μεγαλύτερη πίεση και προωθώντα τη συμμετοχή, την ισότιμη συμμετοχή κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, Υπάρχουν άλλοι ομιλητέ που θα ήθελαν το λόγο. Ε, και εγώ δύο λόγια. Ε, ευχαριστούμε την κυρία Γιακονσάρη. Η κυρία Καστέξ ε, μίλησε για την πρόταση 27 για τις ενδιακές υποδομές. Για μένα είναι ένα οριζόντιο θέμα, γιατί θα πρέπει να συνδεθεί με την, και με την πρόταση 40 που αναφέρεται μια ε, βασική τραπεζική υπηρεσία, μια ελάχιστη τραπεζική υπηρεσία. Χρειάζεται λοιπόν μια ενεργειακή ασπίδα. Ήδη και, και χθε το βράδυ το συζητούσα. Ε, η Κομισιόν έχει την ιδέα να χρησιμοποιήσει την ενεργειακή φορολόγηση, αλλά όχι με στόχο να ε, τεθούν καινούργοι πόροι στη διάθεση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε για να αναδιανεμηθεί κάποιο εισόδημα, όπως γίνεται συνήθως με τη φορολογική πολιτική, αλλά ως τρόπο ε, για την διόρθωση της, ε, του προσανατολισμού της αγοράς. Ποτέ δεν έχει συμβεί αυτό. Ποτέ η φορολογήση δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τέτοιο λόγο στο παρελθόν. Η φορολόγηση χρησιμοποιείται για να αυξηθούν τα έσοδα του κράτους και για να αναδιανεμηθεί το εισόδημα. Πολύ δε περισσότερο που βρισκόμαστε στην περίοδο μετά την κρίση. Με τις ανισότητες να έχουν αυξηθεί σε σχέση με πριν, που υπήρχαν ήδη δηλαδή, τώρα ακόμα περισσότερο. Η ενεργειακή φορολόγηση δεν μπορεί να αγνοήσει την αναδιανομή. Η Κομισιόν ε, προτείνει κατά βάση να γυρίσουμε την πλάτη μας στην κοινωνική δικαιοσύνη. Για μένα χρειάζεται λοιπόν μια ενεργειακή ασπίδα για να συνοδεύσει την μετάβαση προς ένα μοντέλο μικρότερης κατανάλωσης, μικρότερης ενεργειακής κατανάλωσης, που θα επιτρέψει να δοθούν κίνητρα στις αγορές και κίνητρα στους καταναλωτές και σε ό,τι αφορά τη θέρμανση των σπιτιών τους και σε ό,τι αφορά τις μεταφορές για παράδειγμα. Σε ό,τι αφορά τις ε, υπηρεσίες κοινου, ε, ε, γενικού ενδιαφέροντος, η Κομισιόν καθυστερεί στις ε, κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελίας η ευρωπαϊκή, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευρωπαϊκή διάσταση, όχι σε υπηρεσίες όπως η αστυνομία, η δικαιοσύνη κλπ, αλλά σε άλλους τομείς κοινή ωφελία. Για παράδειγμα στις μεταφορές. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, λέω, η ευρωπαϊκή διάσταση αυτών των υπηρεσιών. Όταν υιοθετήσαμε την έκθεση την οποία ήμουν εγώ υπεύθυνη για την κρίση, τι είπαμε πει, τι θα πρέπει να περιμένουμε τον 22ο αιώνα για να σχεδιάσουμε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο σιδηροδρόμων. Πότε θα έχουν πρόσβαση οι ευρωπαίοι καταναλωτές σε ευρωπαϊκές υπηρεσίε μεταφορών. Χρειάζονται υποδομές που θα ενώνουν όχι ίσως τη Βρέστη με το Βλαδιβοστόκ, αλλά τουλάχιστον το Τάλιν με τη Λισαβόνα. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές που θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υποδομέ όμως θα πρέπει να έχουν πρόσβαση και σε μια υπηρεσία κοινή ωφελία σιδηροδρόμων. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να λαμβάνονται οι υπόψη οι επιδοτήσεις. Ε, όταν ξεκίνησε το Θαλής ε, οι επιδοτήσεις που δινόντουσαν στις οικογένειες μέχρι τότε δεν επεκτάθηκαν στο Θαλής γιατί, γιατί το project Θαλής ήταν ένα project ιδιωτικών συμφερόντων υποτίθεται και Ε, θα πρέπει στις καινούργιες υποδομές να έχουν ελάχιστη πρόσβαση μέσω μιας ευρωπαϊκής λογικής και όχι εθνικής λογικής ε, οι όλοι οι καταναλωτές. Τώρα, για την πρόταση 29, κύριε Γιακονσάρη, ε, έχει άποψη. Η Κομισιόν πρέπει να χρησιμοποιεί το άρθρο 9. Σας υποστηρίζω σε αυτό. Και διαπιστώνω ότι η Κομισιόν σκοπεύει να εξετάσει τον κοινωνικό αντίκτυπο όλων, το, όλων των νομοθετικών κειμένων της εσωτερικής αγοράς. Εγώ θα σας πρότεινα να κάνουμε μια λεπτομερή ανάλυση ε, και το προτείνω αυτό κύριε Γιακονσάρη να εξετάσουμε όλες τα νομοθετικά κείμενα που η Κομισιόν έχει εκδώσει από την αρχή αυτής της θητείας της για να δούμε πόσες ε, έχουν συμπεριλάβει ε, εξέταση του αντικτύπου σύμφωνα με το άρθρο 9. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Για την πρόταση 30, η αιώνια συζήτηση με την Κομισιόν που λέει ότι βελτίωση της ε, οδηγίας ε, για τις αποσπάσεις. Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται και σε, μεταξύ μόν, δεν συμφωνούμε μέχρι τώρα, ε, Όμω θα πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία. Ορισμένοι θέλουν αναθεώρηση τη οδηγία και όχι απλώ μια βελτίωση. Θα πρέπει να το δούμε και μεταξύ μα για να αποφασίσουμε. Η Κομισιόν προβλέπει μόνο βελτίωση, όχι αναθεώρηση. Τώρα, πρόταση 32. Ε, βιομηχανικές ε, ε, αναδιαρθρώσεις και πρόβλεψή τους. Θυμάστε το δίκτυο ΙΡΕΝ για την δημιουργία ενός κώδικα δεοντολογίας σε τέτοιου περιπτώσεις αναδιαρθρώσεων. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να εμπνευστούμε από, αυτή την, από, αυτό, το, αυτό το project, το ΙΡΕΝ και τον κώδικα δεοντολογίας που είχε προταθεί πιστεύουμε ότι θα πρέπει να προτείνουμε στην Κομισιόν διάφορα πράγματα που θα ε, λαμβάνονται υπόψη που, ε, έτσι ώστε κάτι της αναδιαρθρώσης να λαμβάνεται υπόψη ο κοινωνικός διάλογος. Τελευταίο σχόλιο για την πρόταση 38, διαχείριση, ε, διακυβέρνηση μάλλον των επιχειρήσεων. Θα πρέπει να μιλήσουμε για την κλίμακα των μισθών, για το μισθολόγιο, ε, για τον περιορισμό των υψηλών ε, εισοδημάτων, για τη θέση ορίου στα ψηλά εισοδήματα, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος ε, η πρόταση που θα υποβληθεί να είναι πολύ ευχάριστη και σεξι, αλλά να μην λύνει τα προβλήματα της διακυβέρνησης. Δηλαδή, θα, μπορούσαμε να, θα μπορούσε να προταθεί ενδεχομένω ε, να προτείνουμε την ε, αύξηση του αριθμού των γυναικών στη, στα ανώτατα κλιμάκια, αλλά αυτό δεν ε, αρκεί για να εξισορροπηθούν ε, τα, τα συμφέροντα της επιχείρησης με τα συμφέροντα των μετόχων. Αυτά. Κύριε Είμαι σίγουρη ότι με βάση τα σχόλια που ακούστηκαν θα μπορέσουμε να ξαναδούμε το κείμενο και να το ε, βελτιώσουμε. Σε ό,τι αφορά τα καινούρια νομοθετικά κείμενα, καταλαβαίνω και συχνά πολλές φορές ε, πετάμε τον μπαλάκι των δικών μας ευθυνών στους ε, ε, νομικούς και στους δικηγόρους. Όπως ξέρετε, είχαμε μια υπόθεση στην Σουηδία μιας απόφασης που ελήφθη από τα δικαστήρια, πολιτική απόφαση όμως κατά βάση. Ε, θα πρέπει να το αποφύγουμε αυτό, τα δικαστήρια να παίρνουν πολιτικές αποφάσεις. Η νομοθεσία λοιπόν θα πρέπει να είναι όσο δυνατόν πιο σαφής γίνεται, γιατί αλλιώς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε αποκτά τον χαρακτήρα κοινοβουλευτική συνέλευση, ιδιαίτερα για κοινωνικά δικαιώματα κλπ. Μην ξεχνάτε ότι ο τίτλο είναι η, Ευρωπαϊκή, η νέα αγορά για τους πολίτες. Η αγορά για τους Ευρωπαίους. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε την ε, νομοπαρασκευαστική διαδικασία με τον τίτλο αυτό ο τίτλος αυτός είναι η αφετηρία θα πρέπει να βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση των πολιτών και νομίζω ότι αυτό θα χρειαστεί ακόμα πολύ προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας όμως. Σας ευχαριστώ. Ναι, το ίδιο χρονοδιάγραμμα ώστε η να μας ακούσει. Λοιπόν, προθεσμία τροπολογιών 26 Ιανουαρίου στις έξι αργά το απόγευμα και πάλι. Άλλη δέσμη τώρα για την οικονομική διαχείριση και εδώ έξι γνωμοδοτήσεις θα πάνε στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή. Έχουμε δύο εισηγητές εκεί, και θα έχουμε κοινή συζήτηση, αυτό σας προτείνω. Ο κ. Καζανγκο ε, για τρία κείμενα, δυστυχώ ε, απόν τώρα, αλλά κυρία Ισαγιά θα λάβει το λόγο που τον αντικαθιστά για το μέρος τουλάχιστον αυτό της συζήτησής μας για αυτά τα τρία με τη σειρά, έτσι. Εδώ πρώτα απ' όλα γιατί πρόκειται για τη μεταβολή του κανονισμού, αλλά και του κανονισμού για τις διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τα υπερβολικά ελλείμματα απαιτήσει που εφαρμόνται στα δημοσιονομικά πλαίσια στα κράτη-μέλη και ακόμα επαγρύπνηση επιθεμάτων προϋπολογισμού στην ε, ζώνη ευρώ. Έχετε το λόγο και μετά θα έχουμε και τις υπόλοιπες τρεις νομοδοτήσεις που είναι μέλος του πακέτου αυτού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, ζητώ συγγνώμη εκ μέρου του Ντέιβιντ που δεν μπορούσε σήμερα να είναι παρόν γιατί ο πρόεδρο Μπούζεκ επισκέπτεται τη Μάλτα και όλοι οι βουλευτέ ε, από τη Μάλτα βρίσκονται εκεί. Εκ μέρου λοιπόν του κ. Κάζα θα παρουσιάσω τι τρει νομοδοτήσει και θα διαβάσω την παρουσίαση που έχει ετοιμάσει ο κ. Κάζα. Καταρχήν, ε, χαίρομαι που μπορώ να σας ενημερώσω ότι και οι δύο εισηγητές για το θέμα αυτό κατάφεραν να έχουν μια κοινή θέση για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε και έχουν ε, μια συντονισμένη θέση, ούτως ώστε να είναι ε, οι προτάσεις τους αρμονικές. Λοιπόν, επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στο ότι θα υπάρχει πάντοτε προσαρμογή στους δημοσιονομικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο στόχο της πρόθεσης, της απασχόλησης και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας παράλληλα με την καταπολέμηση του αποκλεισμού. Δεύτερον, ε, διασφάλιση ότι θα ληφθούν υπόψη ιδιαίτερα τα κοινωνικά θέματα στην παρακολούθηση των κανόνων δημοσιονομικής πειθαρχίας. Τρίτον, διασφαλίζεται ότι τα κονδύλια που συλλέγονται υπό μορφή προστήμων θα χρησιμοποιούνται προ όφελο των μακροπρόθεσμων στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνοχή και δεν θα αναδιανέμονται μεταξύ των συνετών κρατών μελών. Τέταρτον, διασφαλίζεται η ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση. Οι στόχοι τους οποίους μόλις σας διάβασα είναι στοιχεία τα οποία επανέρχονται και στις τρεις εκθέσεις. Θα αναφέρω τώρα τα πιο σημαντικά σημεία αυτών των ε, τριών, γνωμοδοτήσεων. Καταρχήν για τη γνωμοδότηση σχετικά με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Η πρόταση της Επιτροπής θα έπρεπε να αναφέρεται στην κοινωνική διάσταση παράλληλα με την οικονομική διάσταση όταν μιλάμε για τους συνολικούς στόχους αυτού του τομέα. Επιπλέον ε, θα έπρεπε να αναφέρεται ε, η σημασία της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Τέλος, όσον αφορά την εφαρμογή της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες διεξάγονται για να επιτύχουμε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την ανάπτυξη. Περνώ στη δεύτερη γνωμοδότηση τώρα για το δημοσιονομικό πλαίσιο των κρατών μελών. Τα δημοσιονομικά πλαίσια των 100 μελών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων συνταξιοδότησης ε, και ε, περίθαλψη. Και τρίτη γνωμοδότηση για την αποτελεσματική επιβολή της δημοσιονομικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ. Ε, το ισχύον πλαίσιο θα πρέπει σε, περίοδους ύφεσης να επιτυχάνει το στόχο ε, κοινωνική Η πρόταση τη Επιτροπής ε, συμπεριλαμβάνει ένα σύστημα κυρώσεων με το στόχο της ενίσχυσης ε, του προληπτικού και του κατασταλτικού πυλώνα του Συμφώνου σταθερότητα και Ανάπτυξης. Νομίζω ότι θα πρέπει παράλληλα με τις κυρώσεις να διατυπωθεί και ένα σύστημα κινήτρων. Κατά τον τρόπο αυτό θα αναλαμβάνουν την ευθύνη τα κράτη-μέλη και θα ανταμείβονται τα κράτη-μέλη τα οποία επιτυχάνουν πρόοδους. Τέλος, ο κύριος Κάζα μου είπε να σας μεταφέρω ότι περιμένει μια επικοδομητική συζήτηση για τις εκθέσεις του με αρκετές τροπολογίες και το κύριο μήνυμα είναι ότι παρότι αυτό είναι θέμα αρμοδιότητας της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής προς την οποία υποβάλλουμε εμείς τη γνωμοδότησή μας, εμείς θα πρέπει να εστιάσουμε σε θέματα που αφορούν τον τομέα της απασχόλησης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ κύριε Σεία για την παρουσίασή σας και επίσης το ότι σεβαστήκατε τόσο αυτά που απασχολούσαν τον εισηγητή. Ναι. Ε, επιβεβαιώνται όλα αυτά που είπατε εσείς εκ μέρους του κύριου Κάζα και εργαστήκαμε στα πλαίσια μιας καρποφόρου συνεργασίας στο πνεύμα στο οποίο είχε συνεργαστεί και ο κύριο Κάζα ακριβώ όταν για την Οικονομική Νομισματική Επιτροπή είχε συντάξει μια γνωμοδότηση πάνω σε αυτά. Και θα ήθελα μια ελαφρά, ελαφρά μεταβολή της ε, ημερήσιας διάταξης για να στέκουν τα πράγματα συνδυαζόμενα μεταξύ τους. Το σημείο 23 να δούμε που έχει να κάνει με την ίσχυση της εποπτείας δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Εδώ εφόσον πρόκειται βέβαια για το ε, κείμενο το σημαντικότατο, το βασικό για όλο αυτό το σκελετό, το μηχανισμό που γίνεται προσπάθεια διόρθωσης και παράκαμψης των δυσκολιών στην εφαρμογή του σχεδίου σταθερότητας. Τώρα, να σας πω κάτι επίσης εμπειρωματικά που μας απασχολεί και θα ε, δείτε αυτό στις νομοδοτήσεις που σας προτείνουμε. Αυτό το σύνολο της διαχείρισης οικονομικής όπως προτείνει από την Επιτροπή βασίζεται στην νομική Βάση 121 της συνθήκης ε, για το συνδυσμό των οικονομικών πολιτικών που θα πρέπει να θεωρείται σαν ένα θέμα κοινού ενδιαφέροντος ε, και αυτό και για τα κράτη-μέλη της ζώνης ευρώ αλλά και πέρα από αυτήν. Και σε αυτά που μας απασχολούν είναι και το άρθρο 148 να προσθέσουμε για την πολιτική απασχόληση και για τον τρόπο με τον οποίο από κοινού θα πρέπει να ενδιαφέρονται να εργάζονται τα κράτη-μέλη πάνω σε αυτή την πολιτική απασχόληση. Διπλή βάση. Κατά κάποιο τρόπο έχει δεχτεί η Επιτροπή να γίνει έτσι όταν ακριβώς ε, είχε αλλάξει η κατάσταση από τη μια μεριά είχαμε ασχοληθεί με τις διάφορες προσανατολισμούς στους οικονομικούς πολιτικούς και μετά την ε, γραμμή για την απασχόληση και σιγά σιγά με τα χρόνια που πέρασαν φτάσαμε σε αυτή την ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή που βασιζόταν, στηριζόταν σε αυτό το στο διπλό πυλώνα που ήταν μια διπλή πολιτική, την ίδια λογική να θετήσουμε και εδώ, αυτό σας προτείνω διαφορετικά. Το ίδιο το πνεύμα της Συνθήκης Αμφώνας δεν θα γινόταν σεβαστό. Δηλαδή αυτό το άρθρο 9 που θα πρέπει να αποτελεί την γραμμή που θα πρέπει να μας απασχολεί σε αυτήν την κοινωνική πολιτική και με το άρθρο 9, αλλά ταυτόχρονα με αυτή τη διπλή νομική βάση ενδεχόμενα αυτό στην συνθήκη και έτσι ακριβώς κατά την άποψή μου μπορούμε να ενισχύσουμε τον τρόπο αυτό προσέγγισης, το δικό μας δηλαδή. Στην έκθεση για την ενισχύση της εποπτείας και το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Η κυρία Βόρτμαν Κόλ είναι η συγγήτρια στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή. Πέρα από την βάση αυτή την νομική την διπλή, συμπεριλάβαμε και μια έκφραση ανησυχίας ότι σε αυτόν το τομέα η προσέγγιση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της το τι θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, αν αποφασιστεί η στρατηγική του 2020, αν αποφασίζεται, έχουμε μια ενίσχυση των εργαλείων ε, οικονομικής πολιτικής Κάτι που δεν γίνεται έτσι αφηρημένα, αλλά λαμβάνει υπόψη και τη στρατηγική που έχει χαραχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως δεν καταλαβαίνει κανείς τόσο το 2020 την πολιτική στρατηγική στα πλαίσια ενός νομοθετημένου, αλλά θα μπορούσαμε να, να ζητήσουμε η οικονομική αυτή πολιτική να αποφασιστεί, σε συνδυασμό με τους ιδιαίτερους προσανατολισμούς τους συγκεκριμένου με τη γενική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτείνω επίσης ε, παρόμοια ε, ότι να αποφύγει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την προσέγγιση οτιδήποτε ε, θα επαναλάβει αυτή την πολιτική, την οικονομική. Θα πρέπει κανονικά να λάβει υπόψη της και τα ελλείμματα ε, αλλά και τα πλεονάσματα κατά τη διάρκεια του σχετικού κύκλου. Κάτι που σας προτείνω επίσης θα το δείτε να συμπεριλαμβάνετε σε διάφορα σημεία του κειμένου. Στο νόημα αυτό της Επιτροπής πού Putin ε, Fiscal Policy να βάλουμε το αποτελεσματική πολιτική, αυτό το συνετό, τη συνετή πολιτική, γιατί το πρώτο αυτό το συνετή δεν ε, βασίζεται πουθενά συγκεκριμένα, δεν ε, έχει σχέση με μία προσδιορισμένη οικονομική ε, θεωρία είναι κάτι που συμπεριλαμβάνει τώρα εδώ η Επιτροπή σε αυτό και στα πλαίσια που η οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη διπλή πρόκληση δηλαδή τριπλή ίσως και την κρίση αλλά πέρα από την κρίση τώρα και την πρόκληση τη δημογραφική και επίσης την πρόκληση της ανταγωνιστικότητας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό που θα πρέπει να μας επιτρέπει να πετυχαίνουμε οικονομική πολιτική είναι πέρα από τη δηλία, το δισταγμό κλπ. Πρέπει να είναι πάνω απ' όλα η αποτελεσματικότητα. Πρόκειται εδώ για προτάσεις που θα υποβάλει έτσι κι αλλιώς η κυρία Βόρτμαν Κόλ και αυτό στο όλο διατακτικό να συμπεριληφθούν και στοιχεία με αυτό το εξάμενο το ευρωπαϊκό και προτείνω να ληφθούν αυτά υπόψη επίσης γιατί μας αφορούν ιδιαίτερα ε, για να παρακολουθούμε τις κατευθείας γραμμές της απασχόλησης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, νομίζω ότι αδίκως παραμένει σιωπηλή. Αυτό για το πρώτο κείμενο. Έχετε μπροστά σας το σύνολο αυτών των ε, τροπολογιών που προτείνω, αρκετές 62 ε, τροπολογίες, δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω περισσότερο τώρα σε αυτή την παρουσίασή μου. Για τη δεύτερη τώρα γνωμοδότηση που σας παρουσιάζω, στο σημείο 24 γνωμοδότηση για την πρόταση κανονισμού για την πρόληψη και την ρύθμιση της μακροοικονομικής πολιτικής και η Ελίζα Φερέρα είναι στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή σε ηγέτρια. Είναι πολύ σημαντικό και καινοτόμο σε αυτή η δέσμη, γιατί κατά κάποιο τρόπο μέσω της ρύθμισης αυτής προσπαθεί η Επιτροπή να λάβει υπόψη της αυτές τις ελλείψεις που παρατηρούσαμε στην ε, πρώτο αυτό πακέτο διαχείρισης οικονομικής, ε, εντάξει, και τα μακροοικονομικά, να λύσουμε το θέμα με τα μακροοικονομικά στοιχεία αυτών. Και ε, όσον αφορά το νόημα αντιμετωπίζουν προβλήματα σε αυτήν την ομοδότηση, γιατί αυτό όμως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι να αντιγράψουμε απλά και μόνο έτσι σκέτα αυτό το σύμφωνο σταθερότητας, αλλά να δείξουμε μια λογική και έτσι το σύμφωνο σταθερότητας ε, να μπει μέσω συγκεκριμένων δικτών αριθμητικών και όχι μέσω μιας αλληλεπίδρασης ή συζητήσεων ποιοτικών. Για να μπορέσουμε λοιπόν να κατευθύνουμε όπως πρέπει τη στρατηγική των κρατών μελών. Πολύ καλά γνωρίζω ότι με το εξάμεινο το ευρωπαϊκό και με το σχετικό προσδιορισμό σε κάθε χώρα τον Ιούνιο των προσανατολισμών αυτών θα μπορέσουμε να δούμε καλύτερα ειδικότερα την οικονομική πολιτική κάθε κράτους μέλους αλλά ο φόβος μου είναι ότι οι δείκτες οι ποσοτικοί που μας προτείνονται κάπως παρεμποδίζουν την ανάπτυξη μιας εξυπνάδας συλλογική. Ε, και όσον αφορά τα μικροκομμάτια, εντάξει, χαίρομαι τώρα για τη μεθοδολογία να ρωτιέμαι τι γίνεται για τον κίνδυνο να αναπαραχθούν αυτά τα αρνητικά φαινόμενα του Σύμφωνου Σταθερότητας που είχαμε παρατηρήσει. Ένα παράδειγμα, η Ισπανία ήταν η χώρα που το Δεκέμβριο του 2009 ε, για να δω τον Αύγουστο, Αύγουστο, Αύγουστο 2008, αν βάζαμε ένα τριπλό αλφα σε μια χώρα που ανταποκρίνεται στα, ε, στις προϋποθέσεις ακριβώς του συμφώνου σταθερότητας θα ήταν η Ισπανία. Βλέπουμε όμως ότι έτσι δεν εξασφαλιζόταν μια στηρίξιμη ε, και αναπτυσσόμενη έτσι οικονομία. Γι' αυτό λοιπόν και αυτά που είπα για τα μακροοικονομικά. Τώρα για τους ίδιους τους δείκτες ε, που στην πρόταση αυτή θα είναι και το σημείο κλειδί της όλης συζήτησης. Έχουμε και ένα θέμα μεθοδολογίας αλλά και ένα περιεχομένου. Για τη μέθοδο να ε, δω και πάλι την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα έπρεπε να συνδυάσει με τον ορισμό των δικτών αυτών. Από ό,τι μας έχει διδάξει η πείρα, οι δίκτες αυτοί δεν μπορούν να είναι μια, δεν να είναι μια και έξω. Όταν αντιλαμβανόμαστε, οριστική δηλαδή, Τώρα μην ξεκινάμε τώρα με το σύμφωνο σταθερότητο, τι γίνεται, τι δεν γίνεται, γιατί αν είχε εξελιχθεί τότε θα είχαμε καταλάβει τι θα γίνεται, τι γινόταν με τις οικοδομές και, ε, και με όλα αυτά δύσκολα. Εντάξει, εδώ θεωρώ ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, όταν αποφασίστηκε αυτό το Σύμφωνο Σταθερότητα, ε, είχαν την άποψή του που εξέφρασαν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ θα πρέπει να συνεχίσει να συνεργάζεται κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων. Τι σημαίνει ότι οι δείκτες, οι δείκτες για να αποτελούν αντικείμενο τακτικής αναθεώρησης, αυτό θα πρέπει να γίνεται και μετά την αναθεώρηση αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να μπορεί να λέει την άποψή του σχεδόν στην απόφαση και αυτό μέσω της όλης διαδικασίας ε, ανάθεσης ε, αρμοδιοτήτων μέσω του Κοινοβουλίου. Εδώ σχετικά με αυτούς τους δείκτες σας είχα πει λοιπόν ε, ποια θα μπορούσε να είναι ο κατάλογος. Ε, όπω είπαμε πριν και για αυτές τις αρμοδιότητες κατεξουσιοδότηση, και εδώ πρόκειται για μία αντίφαση ίσως. Ε, είναι πολύ ποσοτική και όχι αρκετά ποιοτική. Ταυτόχρονα σας ε, δίνω ένα μακρύ κατάλογο δικτών. Αν έχουμε όμως μια προσέγγιση των δικτών για να έχουμε αυτά τα στοιχεία που να αντιστοιχούν και στις ε, ε, ανησυχίες μας. Ε, σας υποδεικνύω αυτό το κατάλογο που συμπεριλαμβάνει διάφορες προτάσεις που εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα μας απασχολούν στις όλες τις συζητήσεις μας και που κατά την απόψή μου αξίζει να ληφθούν υπόψη και κάθε φορά να έχουμε τη... βλέπουμε ότι χρειάζεται να λαμβάνουμε υπόψη μας την κατάσταση ως έχει ελληματικά ή πλεονασματικά σχετικά με αυτά τα κριτήρια. λοιπόν, γύρω-γύρω από αυτά τα κριτήρια και ακόμα κάτι. Αυτή η προσέγγιση όσον αφορά την ε, έλλειψη ισορροπίας και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έξω από αυτήν. Να πω κάτι ακόμα για τους δείκτες, τους οποίους προτείνω να συμπεριληφθούν όσον αφορά τα φορολογικά κριτήρια. Ήδη το είπα προηγουμένως πάνω σε ένα άλλο θέμα, νομίζω ότι έχει να κάνει με την αρμοδιότητα ακριβώ της Επιτροπής μας. Ο τρόπος με τον οποίο επιβαρύνει τα κεφάλαια ή την εργασία η φορολογική είναι η σημαντική ε, παράγοντες ε, που καθορίζουν ε, την εργασια η ειναι οι σημαντικη παραγοντες που καθοριζουν την ισορροπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το είδαμε πρόσφατα τα θέματα που μας απασχόλησαν σχετικά με αυτούς τους δείκτες τώρα και ένα σημείο που σίγουρα με του συναδέλφου από την Οικονομική Ζωμενική Επιτροπή θα συζητηθεί από κοινού και εδώ να δούμε τι θα γίνει, το ξεκίνημα, πώ μπορεί να είναι γιατί αν λάβουμε υπόψη μα ε, όσα έχουν να κάνουν με τα φορολογικά στην ε, εργασία και στο μια χώρα όπου πάνω σε αυτό επιβάλλεται ιδιαίτερη φορολογία, ενώ αλλού όχι. Εάν οι καλοί δείκτε είναι ε, ο μέσος όρο ανάμεσα αυτά, δεν γίνεται, δεν πάνε τα πράγματα, δεν μπορούν να προχωρήσουν. Έχουμε την κρίση στην αρχή και τώρα πώς γίνεται όλα αυτά τα πράγματα. Το catching up αυτό, τι γίνεται και αυτή την παρακολούθηση ακριβώς για τους καλούς δείκτε. θα έχουμε μια πραγματική δυσκολία που χρειάζεται να ληφθεί υπόψη και να αντιμετωπιστεί. Έτσι, αυτό για την ε, πρόληψη λοιπόν. Για τα μακροοικονομικά, για τα λήψη ισορροπίας δεν θα μακρηγορήσω, θα πρέπει να δώσουμε και χώρο και χρόνο στη συζήτηση και θα δούμε το τελευταίο κείμενο που έχει να κάνει με τις κυρώσεις απέναντι σε αυτές τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Έχει άλλο τίτλο διαφορετικό, μέτρα εκτέλεσης για να ε, λύσουμε προβλήματα παρόμοια μακροοικονομικά στη ζώνη Ευρώπη και είναι έκθεση της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής και την έχει αναλάβει συνάδελφος Καρλ Άγγλουντε. Και στο κείμενο αυτό το σημαντικό έχει να κάνει στα πλαίσια τριών λέξεων, λίγων λέξεων. Πρώτα απ' όλα, δυσκολία να έχουμε μηχανισμούς κυρώσεως που να έχουν να κάνουν μόνο με τα ελλείμματα και όχι τα πλεονάσματα. Δεύτερο, μέσω τη συζήτηση στο Συμβούλιο, στο Μαδεργασία ε, του κ. Ε, Βαμπόη και το, όλες αυτές τις ε, για τα διορθωτικά ελλείμματα και το δικαίωμα ψήφου, όλα αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται στην πρόταση αυτής της Επιτροπής. Οι προτάσεις αυτές θα εξεταστούν όταν κάθε ένα από αυτά τα εργαλεία θα υποβληθεί προς επανεξέταση. Και τώρα στα πλαίσια του προστατισμού του γενικού στα οικονομικά αυτά θα πρέπει να δούμε ποια είναι η απόψή μας, να το εκφράσουμε και τις κυρώσεις ε, για τα θεωρητικά ταμεία και κονδύλια εκεί για τα προβληματικά κράτη θα υπήρχε, θα δημιουργούσαμε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα γιατί είναι κράτη που ξεκινούν από μια άνηση βάση όπου άλλα κρατή διαθέτουν πολλά και άλλα λίγα. και ουσιαστικά θα επιβάλλουμε κυρώσει ε, όσους είναι σε φάση catching up. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι είναι χώρε που ήδη αντιμετωπίζουν έλλειμμα για να... και προσπαθούν να προλάβουν. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να έχουμε κυρώσεις που είναι πραγματικά έξυπνες και αυτή στην ε, συζήτηση αυτού του είδους ε, για το κείμενο αυτό. Τώρα δεύτερο κατά την άποψή μου σημαντικό σημείο είναι ότι αυτές οι κυρώσεις δεν πρέπει να επιβαρύνουν τη γενική στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπω την προσδιορίζουμε, την καθορίζουμε και σε μακροπρόθεσμες φύσεω επενδύσει, όπως παροτρύνουμε. Και ακόμα κάτι τελευταίο, μια συμφωνία και τον κύριο Κάζα. Η πρόταση της Επιτροπής για την αναδιανομή στις καλές θετικές χώρες ποσό αυτών των κυρώσεων δεν νομίζω ότι είναι κάτι θετικό. Αυτές οι έξυπνε κυρώσει που μπορούν να ισχύσουν θα πρέπει ίσως να μπαίνουν στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό για επενδύσεις, χρηματοδότηση επενδύσεων μακροπρόθεσμων και τα ευρωπαϊκά μπόντ και όλα αυτά. Θα δούμε πώς θα ληφθεί η απόφαση. Αυτή την παρουσίαση λοιπόν θα ήθελα να κάνω πάνω σε αυτά τα τρία κείμενα. Με συγχωρείτε, κάπως μακρηγόρησα, συγγνώμη. Τέλο πάντων, προσπάθησα όμω να εκθέσω πλήρω τα πράγματα. Ο κ. Γίγκολτ μου ζήτησε το λόγο. Κάποιο άλλο, μήπω επιθυμεί να λάβει το λόγο επίση. Κρότσμαν. Γίγκολτ. Ε, ευχαριστώ. πολύ για τη δουλειά σας και για το πνεύμα συνεργασίας ε, που σας διακρίνει. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι... έχει ιδιαίτερες ευθύνες για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Το παλιό Σύμφωνο Σταθερότητας και ε, Ανάπτυξης αποφασίστηκε σε μια στιγμή, υιοθετήθηκε σε μια στιγμή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ήταν σύνομοθέτη. Δεν λειτουργήσε σωστά το σύμφωνο αυτό, μεγάλη ανεργία, κοινωνικές ανισότητες στην Ευρωζώνη είναι σημερινά φαινόμενα πλέον, αλλά και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο στην Ευρωζώνη. Τώρα, οι πολίτες αναμένουν μια αναθεώρηση της ε, ε, δομής διακυβέρνησης Ευρωπαϊκή Ένωσης που να δουλεύει. Και αν δούμε τις, ε, την καρδιά των προτάσεων που συζητούμε, τον πυρήνα τους, θα καταλάβουμε ότι στην πραγματικότητα είναι δύο τα βασικά στοιχεία, δύο οι άξονες. Πρώτον, ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και των απαιτήσεων δημοσιονομικής πειθαρχίας και δεύτερον, να προσθεθεί κάτι το οποίο έλειπε στην παλιά δομή διακυβέρνηση οικονομικής διακυβέρνηση και πιο συγκεκριμένα πραγματικές ε, ε, αρμοδιότητες ε, στην οικονομική εξορρόπηση. Όταν δημιουργήθηκε η Ευρωζώνη, οι οικονομικές ανισορροπίες δεν εθίγησαν. Δεν ήταν θέμα εκείνη την εποχή. Το σκεπτικό ήταν, είναι αρκετή δημοσιονομική πειθαρχία. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα όπου η γραμμή σκέψης αυτού του τύπου είναι πολύ ε, ανεπτυγμένη και ισχυρή. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα, υψηλή ανεργία και αυξανόμενες ε, ανισότητες, κυρίως στις χώρες που ήταν οι πιο, δημοσι... Ε, πιο πειθαρχημένες δημοσιονομικά. Κοιτάξτε την Ιρλανδία, κοιτάξτε την Ισπανία. Ήταν οι χώρες οι οποίες πραγματικά ήταν πειθαρχημένες δημοσιονομικά, το πρόβλημά τους ήταν η έλλειψη ισχυρής, ισχυρών κανόνων στην εποπτεία του, του χρηματοπιστωτικού τομέα και ε, χαρακτηρίστηκαν από ε, ε, φούσκες στον ε, τομέα των ακινήτων της οικοδομής. Θα πρέπει λοιπόν να κινηθούμε και προς τις δύο κατευθύνσεις. Σαφέστατα σωστή η δημοσιονομική πειθαρχία ε, διότι είδαμε ποια τα προβλήματα σε χώρες όπως η Ελλάδα, παρόλο που σε μεγάλο βαθμό και εκεί το πρόβλημα προερχόταν από την αύξηση του ιδιωτικού χρέους και όχι τόσο του δημοσίου, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν δείτε τις ε, προτάσεις, δεν είναι ισορροπημένες, ε, δεν θα δουλέψουν στην πράξη αν δεν τροποποιηθούν. Γι' αυτό το λόγο το Κοινοβούλιο έχει βαριά ευθύνη Ξέρουμε πώς λειτουργεί το Συμβούλιο. Κάθε κράτος μέλος θέλει να προστατεύσει τους δικούς του οικονομικούς εθνικισμούς. Και το Συμβούλιο δεν μπορεί να δουλέψει με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό το λόγο το Κοινοβούλιο πρέπει να δράσει υπέρ του κοινού ευρωπαϊκού ωφέλους και όχι υπέρ του α ή του β οικονομικού εθνικισμού. Να σας πω ποιε είναι οι βασικέ αδυναμίε τη πρόταση. Και η δική μα Επιτροπή έχει σημαντικό ρόλο διότι αν δεν λειτουργήσει και το κοινωνικό σύστημα θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο η ενεργεία και οι κοινωνικέ ανισότητε. Λοιπόν, οι αδυναμίε, τι δεν θα δουλέψει. Είπαμε, η δημοσιονομική πειθαρχία είναι απαραίτητη. Ακόμα και πιο ισχυρή δημοσιονομική πειθαρχία. Όμω, αν δεν λαμβάνει υπόψη του επιχειρηματικού κύκλου ή του κύκλου οικονομία, τελικά θα η πειθαρχία αυτή θα οδηγήσει σε υψηλότερο χρέος και υψηλότερη ενεργεία. Ε, συνεπώς η δημοσιονομική ε, πειθαρχία δεν μπορεί να είναι αυτόματη. Ε, η πρόταση της Κομισιόν δεν έχει οικονομική βάση. Δεύτερον, η πρόταση ε, επιμένει ιδιαίτερα στην πειθαρχία σε ό,τι αφορά τα έξοδα, στο σκέλος των εξόδων. Όμως δεν μιλάει για το σκέλος των εσόδων, γιατί τα έσοδα είναι πρόβλημα. Τα κράτη-μέλη ακόμα ε, υφίστανται την το φορολογικό ανταγωνισμό. Ε, καταλαβαίνω ότι ε, είναι δύσκολο να υποβάλει κανεί προτάσει για ελάχιστη φορολογία κλπ. Και ενδεχομένως ε, θα μπορούσε κανείς να πει ότι τεχνικά δεν, δεν εντάσσεται αυτή η πτυχή στη συγκεκριμένη έκθεση, αλλά πολιτικά εντάσσεται. Τρίτο, τρίτη αδυναμία, ε, το βαθμονόμιο. Θα μπορούσε κανείς να πει, αν βάλει κανείς πολλά κριτήρια στο βαθμονόμιο για τις ε, θα γίνει το σύστημα λίγο δύσχριστο. Όμως, αν δεν βάλουμε όλα τα απαραίτητα κριτήρια, τα βαθμονόμια δεν θα λειτουργήσουν. Κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, παράδειγμα, είναι σημαντικά. Επίσης υπάρχει και άλλο ένα θέμα, το οποίο είναι επίμαχο στο Συμβούλιο και ασαφές στην πρόταση Κομισιόν. Θα πρέπει να μιλάμε μόνο για τις χώρες με ελλείμματα και για τις χώρες με πλεονάσματα. Ε, είναι θέμα λογικής. τα αίτια για ανισορροπίες ε, στη χώρα της Ευρωζώνης μπορεί να είναι ε, να οφείλονται σε πλέον ελλείμματα, αλλά μπορεί να οφείλονται και σε πλεονάσματα. Για παράδειγμα, μια χώρα η οποία δεν αυξάνει τους μισθούς, ε, είναι εύκολο να δημιουργήσει, είναι πιο εύκολο να δημιουργήσει πλεονάσματα, εμπορικά πλεονάσματα, από ότι μια χώρα που αυξάνει τους μισθούς, ε, με τη μαριθμική αναπροσαρμογή. Είναι προφανές λοιπόν ότι το πλεόνασμα μιας χώρας μπορεί να δημιουργήσει έλλειμμα σε μια άλλη. Γι' αυτό το λόγο η Κομισιόν θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις πραγματικές αιτίες των ανισορροπιών και στα ελλείμματα αλλά και στα πλεονάσματα. Και δεν είναι αρκετό να επιβάλλουμε αυστηρότερες κυρώσεις στις χώρες που ε, αντιμετωπίζουν προβλήματα. Θα πρέπει να υιοθετήσουμε και κίνητρα, μέτρα δηλαδή που θα βοηθήσουν τις χώρες να βγουν από τα δεινά τους, πολιτικές και προσεγγίσεις που θα βοηθήσουν τις διάφορες χώρες να επανέλθουν στον οικονομικό δυναμισμό. Γιατί αλλιώς τα μέτρα αυτά θα καταλήξουν σε μεγαλύτερο έλλειμμα. Τέλος, το είπε και η Περβόνς, θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ καλά τις προτάσεις αυτές που περιμένουμε, γιατί σε μεγάλο βαθμό οι προτάσεις κομισιών αντικατοπτρίζουν το εξή σκεπτικό. Έχουμε ένα νόμισμα αλλά δεν διαθέτουμε ε, μια πραγματική πολιτική ένωση. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να επιβάλλουμε πολύ αυστηρούς κανόνες που θα λειτουργούν πιο αυτόματα. Ακριβώς διότι δεν έχουμε μια δομή η οποία να παρομοιάζει με, την, με μια κυβέρνηση και μπορεί να πάρει έξυπνες ε, αποφάσεις. Ε, όμως, τα πράγματα είναι πολύ περίπλοκα και ο αυτοματισμός ε, δυσχεραίνει τις καταστάσεις. Η οικονομική κατάσταση είναι περίπλοκη και ρευστή. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα-δύο κανόνες μόνο. Συνεπώς, ε, Πιστεύω ότι στην Ευρωζώνη χρειαζόμαστε μια πραγματική οικονομική ένωση που θα έχει εξουσίες να παίρνει αποφάσεις που θα είναι πιο ευφυής από ένα απλό αυτόματο μηχανισμό. Ε, μια, ένας μηχανισμός, ε, μια διαδικασία η οποία θα λαμβάνει υπόψη όλους τους απαραίτητους παράγοντες. Μια, ένα αυτόματο σύστημα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αυτά θα υποβάλουμε τροπολογίες και βέβαια θα υποστηρίξουμε σε μεγάλο βαθμό πολλά από αυτά τα οποία είπατε κι εσείς. Τελειώντας να πω, να επαναλάβω ότι έχουμε ένα, ένα ε, βαρύ φορτίο αν θέλουμε να παίξουμε ρόλο στην ε, ανάπτυξη και την εμβάθυνση του ευρωπαϊκού project ολοκλήρωσης. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να παίξουμε σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ιδιαίτερα η Επιτροπή Απασχόλησης ε, μπορεί να ε, κινητοποιήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, για να πολεμήσει για την μείωση των ανισοτήτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαιρετίζουμε την πρόταση της Επιτροπής γιατί αποτελεί σημαντική συνεισφορά για την ε, αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς το κοινό νόμισμα. Ε, το προτινόμενο σύστημα ε, κυρώσεων που αποτελείται από το τοκοφόρους και μη τοκοφόρους καταθέσεις είναι μόνο ένα βήμα στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος θα πρέπει να προσέξουμε τη διαφοροποίηση. Το σύστημα κυρώσεων θα πρέπει να διευρυνθεί ούτως ώστε ε, ε, να μην διατίθενται προς το κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται ε, χρήματα από, τον τα κοινοτικά διαρθρωτικά ταμεία όσον αφορά την αντίστροφη ψηφοφορία στο Συμβούλιο, νομίζω ότι είναι ένα σύστημα το οποίο πρέπει να διατηρηθεί ως πρόταση. Επίσης, το δημοσιονομικό πλαίσιο για τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι δεσμευτικό η πολιτική Ευρώπη, η στρατηγική Ευρώπη 2020 θα πρέπει να είναι κατευθυντήρια γραμμή μας, θα πρέπει να είναι ένα σημαντικό εργαλείο που θα μας καθοδηγεί στους στόχους ε, στρατηγικής 2020 θα πρέπει να συνεισφέρει και το τωρινό πακέτο για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών. Και η χρήση αυτού του πίνακα βαθμολογίας από την Επιτροπή θα βοηθήσει να κατευθυνθούμε προς αυτό το στόχο. Χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο το οποίο θα αποτελέσει ένα μέσο προστασίας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 ε, τα κράτη-μέλη που δεν μπορούν να πάρουν πιστώσεις από την αγορά θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν από αυτό το νομισματικό ταμείο και θα πρέπει να υπάρχει ως προϋπόθεση το να έχει καταστρώσει ε, το εν λόγω κράτος μέλος ένα πρόγραμμα σύμφωνα με τις συστάσεις του, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ε, και της Επιτροπής. Διαφορετικά θα πρέπει να ισχύσει μια διαδικασία ε, ε, υπερβολικού ελλείμματος ε, με όλες τις διατάξεις που αφορούν την μη φερεγγιότητα. Αυτές είναι οι βασικές μου παρατηρήσεις και νομίζω ότι στο πλαίσιο της συζήτηση μπορεί να προκύψουν και κάποια περαιτέρω θέματα προς συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κοφεράτη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σίγουρα όταν τα θέματα αυτά είναι περίπλοκα και λόγω της περιπλοκότητας αυτής ε, βλέπουμε ότι χωρίζονται σε διάφορες ενότητες προτάσεων διαφορετικών εργασίας. Ε, πάντα έχουμε το πρόβλημα του συνδυασμού ανάμεσα στο ένα και στο άλλο και τη συνοχή τους ανάμεσα αυτό που αποφασίζεται πάνω σε ένα σημείο και τη γενική εικόνα με το γενικό πλαίσιο που θα πρέπει να ισχύει. Ιδιαίτερα κατανοώ και εκτιμώ και τον μόχθο σας το θέμα αυτό της συνοχής της έκθεσης με τις προτεραιότητες των πολιτικών οι οποίες και συμπεριλαμβάνονται στην πρόταση για την ε, Ευρώπη του 2020 πάνω σε αυτά χρειάζεται να κοιτάξουμε με ιδιαίτερη προσοχή. Να σας πω ένα παράδειγμα και στην υπόλοιπη συζήτηση θα μπορούσαμε να επανέλθουμε πάνω σε πολλά και διάφορα θέματα. Το είπαμε, επαναλάβαμε ότι είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να πρικοδοτηθεί με αυτόνομο προϋπολογισμό, να έχει τους πόρους της και να προέλθουν από τα Eurobonds ε, είτε και μαζί με φορολογία πάνω στις ε, δημοσιονομικές συναλλαγές και το συζητήσαμε και ιδιαίτερα έντονα και στο Συμβούλιο για να δούμε και τι γίνεται με τον απροσδιορισμό του προϋπολογισμού αυστηρού πέρα από τις διαθέσεις των κρατών μελών ο γενικός μας πρωτοανστατολισμός, αυτή η δημοσιονομική αυτονομία και για τη διάθεση των πόρων που θα πρέπει και να εξυπηρετούν και για την αντιμετώπιση των κρίσεων, αλλά και για τη στήριξη των πολιτικών ανάπτυξης. Αυτά άμεσα μας βάζουν στη θέση να ψάχνουμε για αυτή τη συνοχή για την οποία αναφέρθηκα πάνω σε ένα κυρίως μεγάλο θέμα, τις αλλαγές στο Σύμφωνο Ανάπτυξης Σταθερότητας. Αρκετά συχνά συζητήσαμε και άκουσα και σήμερα να επαναλάβανε τη ίδια συζήτηση για τη δυνατότητα ενός συστήματος κυρώσεων όπως προβλέπετε και όπως επίσης και ένα σύστημα παροτρήσεων, κινήτρων. Εδώ δεν με πείθουν τα πράγματα. Καταλαβαίνω το λόγο για τις κυρώσεις. Νομίζω ότι συνάδει με την παρότρινση για ενάρετες πράξεις που θα σέβονται τους κανόνες, αλλά δεν καταλαβαίνω αυτό τα, αυτά τα περιπαροτρήσεων, κινήτρων γιατί ίσως διατρέξουμε ένα κίνδυνο να ευνοήσουμε ορισμένα κράτη μόνο και μόνο επειδή δέχονται, σεβόνται τις ρυθμίσεις. Δηλαδή να επιβραβεύουμε όποιον κάνει σωστά τη δουλειά του. Τότε μπαίνουμε σε μια κάπως επικίνδυνη φάση διάσταση δεν υπάρχει πια ενδιάμεσος χώρος. Ε, δηλαδή αυτό το κανονικό, τι γίνεται, τι είναι. Όποιον δεν σέβεται να τον τιμωρούμε. Αλλά τον επιβραβεύουμε όποιον τον σέβεται, αυτό δεν στέκει κατά την απόψή μου. Και να προσθέσουμε και άλλη μια απόψη για να ασχοληθούμε με αυτή την ειδική πτυχή περί κλπ. Εδώ για τις κυρώσεις και για τις νομισματικές επιπτώσεις από αυτές τις κυρώσεις. Αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν παρά μόνο για να ενισχύσουν την αυτονομία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν όλα αυτά να πάνε σε επενδύσεις. Εάν με διαφορετικό τρόπο θέλαμε να τα χρησιμοποιήσουμε να στραφούν αλλού, τότε θα οξύναμε τις αντιφάσεις, αντιθέσεις που λέμε ότι θέλουμε να παρακάμψουμε και να λύσουμε θα μπορούσα να πω και άλλα πράγματα. Εντάξει, μη μακρηγορήσω τώρα. Αλλά σημαντικότατο είναι κάτι την απόψή μου να έχουμε και μια γενική άποψη του ολοπλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης τον ειδικό χαρακτήρα των ενεργειών που ενισχύουν αυτή την ε, εικόνα, αυτό το πλαίσιο και να μην έχουμε αντιφάσεις καινούριε που θα δημιουργήσουν εντάσεις και ρήξη σωστών σχέσεων ανάμεσα στις ίδιες τις χώρες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητάει κανεί άλλο το λόγο. Θα δώσω λοιπόν στην ε, κυρία Έλληνα Φλόρε το λόγο εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι στο παρόν στάδιο δεν είναι κατάλληλη στιγμή για να συζητήσουμε σε βάθος πολλές από τις νέες ιδέες που βρίσκονται στις εκθέσεις σας. Θα περιοριστώ λοιπόν σε πέντε σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτον, θέλω να ευχαριστήσω τους συζητητές και όλους τους συμμετέχοντες για τη συζήτηση. Νομίζω ότι ε, στην ε, έκθεση υπάρχει προσπάθεια συνοχής με την προσπάθεια της Επιτροπής και με την έκθεση της Επιτροπής ε, Οικονομικών Υποθέσεων. Άρα νομίζω ότι είναι καλή βάση για την περαιτέρω συνέχιση των εργασιών. Υπάρχουν ενδιαφέρουσες ιδέες στην έκθεση που θα τις εξετάσουμε στη συνέχιση της συζήτησης. Δεύτερον, ε, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το νομοθετικό πακέτο δεν είναι το παν, δεν είναι η πλήρης απάντηση. Αυτά τα έξι νομοθετικά κείμενα αποτελούν τμήμα της απάντησης. Υπάρχουν πολλά στοιχεία λοιπόν. Εδώ συζητάμε μια συνεκτική απάντηση προς την κρίση. Θα δείτε ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία, αλλά υπάρχουν ε, διάφορες ε, μελλοντικές εξελίξεις. Ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο χρηματοπιστωτική σταθερότητα κλπ. Και υπάρχει και ένα πακέτο διαρθρωτικών μέσων, όπως θα τα αποκαλούσα, που είναι μέτρα πολιτικές που πρέπει να λάβουν τα κράτη-μέλη για να ενεργοποιήσουν το δυναμικό ανάπτυξης που έχουν. Μαζί με τα μέτρα αύξησης της ανάπτυξης που πρέπει να υποστηρίζουν τις εθνικές διαρθρωτικές πολιτικές. Υπάρχει λοιπόν μια ολόκληρη δέσμη μέτρων πολιτικής και αυτό ελπίζουμε ότι θα έχουμε στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης εποπτείας, ούτως ώστε να υπάρχει συνοχή μεταξύ όλων των τμήματων αυτής της δέσμης μέτρων. Αυτά τα έξι νομοθετικά κείμενα δεν θα πρέπει λοιπόν να τα θεωρήσετε ως το μόνο που κάνουμε για να ανταποκριθούμε σε αυτά που χρειάζονται για να βελτιώσουμε την οικονομική διακυβέρνηση. Τρίτο σχόλιο. Είναι πιο συγκεκριμένο, αλλά νομίζω ότι προχωρεί και λίγο περισσότερο αφορά το θέμα των κυρώσεων και του πίνακα βαθμολογίας και των δικτών. Θέλουμε να ενισχύσουμε τη δυνατότητα εφαρμογής της νομοθεσίας και υπάρχει και ένα είδος αυτοματισμού εδώ, αλλά ιδίως ο πίνακας βαθμολογίας παίζει το ρόλο του ότι θα αποτελέσει το έναυσμα εμπεριστατωμένη συζήτηση. Μπορεί να πείτε ότι δεν χρειαζόμαστε ένα πίνακα βαθμολογία για να το κάνουμε αυτό, αλλά κρίνοντα από την εμπειρία μα, βλέπουμε ότι αυτή η εμπεριστατωμένη συζήτηση δεν λαμβάνει χώρα. Ανέφερε η πρόεδρο κάποια παραδείγματα από το παρελθόν, κάποιε χώρε που είχαν πολύ καλή δημοσιονομική κατάσταση, αλλά ξέραμε ότι δεν ήταν επαρκή η μακροοικονομική του ισορροπία. Αν είχαμε αυτή την νομοθεσία, θα είχε γίνει μια εμπεριστατωμένη ανάλυση. Αυτό για να δώσω μια εικόνα του τι μπορούμε να επιτύχουμε με αυτά τα μέσα που προτείνονται. Τέλος, θέλω να τονίσω ότι αν εγκρίνουμε αυτό το νομοθετικό πακέτο εγκαίρως, θα λάβουμε θα κάνουμε ένα βήμα για να ενισχύσουμε την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών αρχών. Θα δείξουμε ότι μπορούμε να λαμβάνουμε εγκαίρως μέτρα, ούτως ώστε να εφαρμόζονται αυτά τα οποία απαιτούνται. Η Επιτροπή λοιπόν είναι πρόθυμη να βοηθήσει, όπως κάναμε και μέχρι τώρα. Είμαστε πρόθυμοι να συνεχίσουμε τις συζητήσεις και θα συνεχίζουμε να παίζουμε το ρόλο μας ούτω ώστε να βελτιωθεί η αξιοπιστία ε, της δυνατότητάς μας να λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σαϊά. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας και θα τα μεταφέρω στον κύριο Κάζα. Θα ήθελα εδώ να δώσω την προσωπική μου απάντηση τώρα, κυρία Κοφεράτη, σε αυτό που είπατε ότι δεν συμφωνείτε με την ιδέα του να επιβραβεύσουμε αυτούς που ακολουθούν τους κανόνες. Προσωπικά συμφωνώ μαζί σας, γιατί οι αγορές επιβραβεύουν αυτούς ε, που τα πάνε καλά και δίνουν βαθμολογία τριπλού α σε αυτούς που ακολουθούν τους κανόνες και βάζουν σε χειρότερη βαθμολογία αυτούς που δεν ακολουθούν τους κανόνες. Αυτό μόνο ήθελα να πω εγώ ως δική μου παρατήρηση. Θα μεταφέρω τα σχόλια στον κύριο Κάζα. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Δύο παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω. Πρώτον, ε, για το πώς λαμβάνεται υπόψη η χρηματοδότηση των ε, συνταξιοδοτικών ε, συστημάτων. Στη μεταρρύθμιση του πακέτου του Συμφώνου Σταθερότητας το 2005 είχα πει ότι αν στους μηχανισμούς του Συμφώνου Σταθερότητας υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μία πρημοδότηση για τις χώρες που θεσπίζουν ένα σύστημα χρηματοδότησης ε, των συντάξεων κεφαλαιοποιητικό, υπάρχει άμεση παρέμβαση των Βρυξελών στη συζήτηση που διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο. πάνω σε βασικά στοιχεία της κοινωνικής συνοχής. Και αφετέρου, υπάρχει μια ανισορροπία όσον αφορά τη συνοχή. Η κυρία Φλόρες είπε ότι έχουμε μια συνεκτική προσέγγιση. Να, είμαστε, να δείξουμε συνοχή λοιπόν μέχρι τέλους. Και αν είμαστε μέχρι τέλους ε, συνεπείς θα πρέπει να έχουμε μια ευρεία αντιμετώπιση και να λαμβάνουμε υπόψη όλα τα στοιχεία που υπάρχουν επιτάπητος. Και μεταξύ όλων αυτών των στοιχείων Υπάρχει κάτι που πρέπει τώρα να το λάβουμε υπόψη μας και είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 και αυτή η στρατηγική απαιτεί μακροπρόθεσμες επενδύσεις που κάπως πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Και αν προσπαθούμε να καθορίσουμε προτεραιότητες, θα πρέπει να δούμε τις δαπάνες που χρειάζονται τα κράτη-μέλη για ένα συνταξιοδοτικό σύστημα κεφαλαιοποιητικό και θα πρέπει να δούμε τις επιπτώσεις ε, στις, τις μακροπρόθεσμες ε, αυτών των επενδύσεων. Ε, ξέρω ότι είναι δύσκολο το θέμα γιατί και βρισκόμαστε μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναδιάρθρωσης παγκοσμίω. Τώρα, κάποιες άλλες παρατηρήσεις για την έκθεση για την οποία είναι αρμόδιος ο κ. Κάζα για το δημοσιονομικό πλαίσιο των κρατών μελών. Ξέρω ότι αυτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέκυψε από την όλη συζήτηση για την ποιότητα των στατιστικών δεδομένων και για την αναγκαιότητα να έχουν τα κράτη-μέλη σωστά μέσα κατεύθυνση των πολιτικών τους. Εποφελούμεθα της ευκαιρίας αυτής. Ε, λέμε να έχουν, ότι θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τα κατάλληλα μέσα καθοδήγησης των πολιτικών. Αυτό το οποίο μας λείπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ότι δεν φαίνεται πώς συνεισφέρουν οι προϋπολογισμοί των κρατών μελών με ποιοτικό τρόπο στην υλοποίηση των στρατηγικών που αποφασίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Στη στρατηγική 2020 υπάρχει ένας μακροπρόθεσμος στόχος καταπολέμησης της φτώχειας. Δεν υπάρχει όμως όραμα για την ποιότητα των δαπανών των κρατών μελών ή έστω και για το ύψος των δαπανών των κρατών μελών προς την προτεραιότητα αυτή. Το μόνο κριτήριο είναι το κριτήριο του Συμφώνου Σταθερότητας, δηλαδή το έλλειμμα μέχρι τώρα και το χρέος. Και όπως είπε ένας πρώην πρόεδρος της Επιτροπής, είναι ανόητα τα νούμερα αυτά. εξετάζουμε τις κατευθυντήριες γραμμές για τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών. Θα πρέπει λοιπόν το δημοσιονομικό αυτό πλαίσιο ε, να επιτρέπει να βλέπουμε ποια είναι η συνεισφορά των προϋπολογισμών των κρατών μελών ε, στους προσανατολισμούς της στρατηγικής του 2020 και ξέρω ότι και ο πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών συμφωνεί με αυτή την ανάλυση. Όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση, μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι στον πυρήνα των μελημάτων μας, αλλά είναι κάπως δευτερογενές. Πάντως πιστεύω ότι πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Όσον αφορά αυτό που είπε η κυρία Έλενα Φλόρες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ναι, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά ε, που έχουν ε, μείνει κατά μέρο στη συζήτηση αυτή και πρέπει να ληφθούν υπόψη. Με βάση αυτά που συζητούνται και αλλού για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, παραδείγματο χάρη, ή για την Στρατηγική 2020, ή και για την αναθεώρηση της συνθήκης ενδεχομένω. Νομίζω ότι πρέπει όλα αυτά να τα έχουμε κατά νου όταν συζητάμε αυτό το θέμα. Σα ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σα στη συζήτηση. Πιστεύω ότι ήταν χρήσιμη η συνεισφορά σα για όλους. Για να δράσουμε εγκαίρως για τη συζήτηση στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή, θα πρέπει να έχουμε ως το δυνατόν υψηλότερη πλειοψηφία για το πακέτο αυτό και να φτάσουμε έγκαιρα και στη συζήτηση στο Συμβούλιο. Γι' αυτό έχουμε βάλει προθεσμία για τις τροπολογίες 4 Φεβρουαρίου το μεσημέρι και θέλουμε να ψηφίσουμε στις 16 Μαρτίου. Θα μας μείνει μια μέρα για τις διαπραγματεύσεις. Και η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να ψηφίσει στις 19-20 Απριλίου, ούτω ώστε να συζητηθεί, να εξεταστεί αυτό το θέμα τον Ιούνιο. Αυτά λοιπόν για τις πρωινές μας εργασίες. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας στην πρωινή συνεδρίαση και θα τα ξαναπούμε στις 3. Θα κάνουμε ανταλλαγή απόψεων με την Ουγγρική Προεδρία.